Συνάδελφοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ παρά τις αλλαγές που έγιναν στην σε διάταξη και τη σειρά με την οποία θα συζητηθούν τα θέματα. Ξεκινάμε λοιπόν ε, λίγο νωρίτερα από τη συνήθως. Επόμενο σημείο που θα συζητήσουμε είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον υποστράτηγο Πασκάλ Σιφολό, διοικητή της Ευρωπαϊκής Διοίκησης Αεροπορικών Μεταφορών, μέδρα του Αιντχόφεν, που ιδρύθηκε το 2010, αν δεν κάνω λάθος, και που έχει αναπτύξει τις ε, επιχειρησιακές της ικανότητες. Θεωρείται ως ε, μια επιτυχής ιστορία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Έχουμε ήδη παρακολουθήσει μια σειρά από παρουσιάσει σήμερα. Είχαμε μαζί μας τον πρόεδρο της Στρατιωτική Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υψηλό βαθμό της βουλγαρικής κυβέρνησης. Καθώς και ένα πάνελ για την στρατιωτική κινητικότητα με την οποία και την πρωινή μας συνεδρίαση όπου συμμετείχαν πέντε πολύ σημαντικοί ομιλητές που μας παρουσιάσαν τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις τους από την σκοπιά του ο καθένας. Είχαμε μαζί μας εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, της ΕΙΕΔ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά το ΝΑΤΟ. Με θέμα, όπως είπα, τη στρατηγική κινητικότητα. Μαζί μας είχαμε τον Διευθυντή Μαρτή, αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Ικανοτήτων Εξοπλισμού Τεχνολογίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, Και τώρα έχουμε μαζί μας τον διοικητή της Ευρωπαϊκής Διοίκησης Αεροπαρικών Μεταφορών που θα μας μιλήσει μεταξύ άλλων και για το θέμα της ε, στρατιωτικής κινητικότητας. Χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, να δώσω λοιπόν το λόγο στον υποστράτηγο Πασκάλ Σιφόλο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την εισαγωγή. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, ως διοικητής της EATC είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα το απόγευμα για να προσπαθήσω να σας εξηγήσω τι είναι η Ευρωπαϊκή Διοίκηση Εναέριων Μεταφορών, πώς λειτουργεί και όπως ανέφερε και η Πρόεδρος γιατί θεωρείτε ότι η διοίκηση μας έχει στεφτεί με επιτυχία θα σας δώσω Κάποιου βασικούς λόγους, αν μου επιτρέπετε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η ιδέα για μια Ευρωπαϊκή Μονάδα Εναέριων Μεταφορών γεννήθηκε στα τέλη του τελευταίου αιώνα με μια διμερή πρωτοβουλία Γερμανίας και Γαλλίας και βλέπετε εδώ στη διαφάνεια ότι χρειάστηκαν περίπου 10 χρόνια για να οριμάσει η σκέψη αυτή, για να καθοριστούν οι λεπτομέρειες, να, δημιουργηθεί, να θεσπιστεί ένας κοινό ε, κανονισμός, να βρεθούν οι τρόποι προκειμένου να ε, καθοριστούν οι κανόνες μεταξύ των τεσσάρων χωρών ιδρυτών αυτή τη διοίκηση και τελικά καταλήξαμε το Σεπτέμβριο του 2010 στην ίδρυση αυτή τη διοίκηση. Μετά από δύο χρόνια προσχώρησε το Νοέμβριο του 2012 συγκεκριμένα το Λουξεμβούργο και έπειτα από άλλα δύο χρόνια περίπου, τον Ιούλιο του 2014 είχαμε την προσχώρηση της Ισπανίας ενώ το Δεκέμβριο του 2004 προσχώρησε και η Ιταλία στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση ενέργων Μεταφορών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε 7 έθνη, μία διοίκηση, μία επιχειρησιακή διοίκηση και επιμένω σε αυτό γιατί είμαστε επιχειρησιακή μονάδα, ε, λειτουργική και επιχειρησιακή επί 24 ε, ώρου βάσεως με 215 μέλη του προσωπικού. Αυτή η διαφάνεια είναι και η πιο σημαντική της παρουσίασης. Σας παρουσιάζω εδώ το επιχειρησιακό μας μοντέλο. Αριστερά βλέπετε τους τρεις βασικούς τομείς ε, δράσης και εμπειρογνωμοσύνης μας, ενάεριες μεταφορές, εναέριος ανεφοδιασμός καυσίμων και αεροιατρική εκένωση. Βλέπετε εδώ ε, στη μέση τον οργανωτικό, το οργανόγραμμα ε, του, του EATC. Έχουμε έναν επιχειρησιακό πυλώνα και έναν λειτουργικό πυλώνα που υποστηρίζει τις βασικές μας ε, ε, δραστηριότητες, ενώ έχουμε και σχέσεις με εξωτερικές ε, οργανώσεις και χώρες και με όλα τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας καταρτίζουμε και χαράσουμε τα σχέδιά μας για το μέλλον. Λαμβάνουμε λοιπόν αιτήματα εναέρειας μεταφοράς από ένα από τα κράτη-μέλη της διοίκησης. Στη συνέχεια Υπάρχει ο σχεδιασμός, η ανάθεση καθηκόντων, ο έλεγχος των ε, επιχειρήσεων, ανάλυση υποβολή εκθέσεων που είναι το τελευταίο βήμα. Ταυτόχρονα όμως λειτουργεί και ο λειτουργικός πυλώνας, ε, ο οποίος τροφοδοτεί τον επιχειρησιακό πυλώνα μέσω των κοινών κανόνων, μέσω της διεξαγωγής μελετών, ε, εποφελία των συμμετεχουσών χωρών και μέσω της εναρμόνισης αλλά και της αύξησης και της ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων μας. Διαλειτουργικότητα σημαίνει στις ένοπλες δυνάμεις να μπορούν, ένοπλες δυνάμεις, να μπορούν να συνεργάζονται στο πεδίο της μάχης. Δεξιά βλέπετε τις ε, συμμετέχουσες χώρες. Είναι κάποιες από τις δεσμεύσεις τους, τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματα. Πρώτον, Όταν μια χώρα προσχωρεί στο EATC, μεταφέρει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμεύουν στον ανεφοδιασμό ε, από αέρος. Αλλά κάρτ, ό,τι θέλουν. Οι τρεις χώρες ε, ε της, ε, της για παράδειγμα, έχουν δώσει το σύνολο των σχετικών τους υποδομών στην EATC. Δεν ισχύει αυτό όμως για όλες τις χώρες. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ε, ανάκλησης, μεταφοράς ε, εξουσίας, χωρίς μάλιστα αναφορά λόγου, χωρίς αιτιολόγηση. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να το κάνει αυτό μια χώρα. Είναι εγγύηση της εθνικής κυριαρχίας και αυτό. Υπάρχει και ένα εικονικό νόμισμα, το οποίο χρησιμοποιούμε. Δεν έχουμε ε, ροές κεφαλαίου, ρευστού, ε, στο πλαίσιο της EATC χρησιμοποιούμε την τεχνική συμφωνία για, την, για τις μεταφορές, τον εναέριο ανεφοδιασμό και τις ανταλλαγές υπηρεσιών, ατάρες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να μπορεί μία χώρα να χρησιμοποιεί ένα περιουσιακό στοιχείο άλλης χώρας μέσω ε, του συστήματος. υπάρχει μια συγκεκριμένη αποτίμηση δηλαδή σε αυτό το εικονικό νόμισμα της χρήσης συγκεκριμένων ε, πόρων ε, της κάθε χώρας. Ε, αυτό το σύστημα δημιουργήθηκε στις ε, αρχές του 2000. Συμμετέχουν και άλλες χώρες, όχι μόνο ευρωπαϊκές, και η ΕΠΑ και ο Καναδάς και ε, ε, αφορά τα MCCE, ε, την, τη συνοδευτική δηλαδή συμφωνία στο Ατάρις. Αυτή η, αυτή η διάταξη, αυτή η διευθέτηση αφορά και ε, την, τις εθνικές δομές της διοίκησης των ε, στρατευμάτων. Γι' αυτό και ε, στις ενέργειες μεταφορές είμαστε πλήρως ενταγμένοι ε, στο σύστημα των επιμέρους χωρών. Και τέλος υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο που εξασφαλίζει την εθνική κυριαρχία. Όπως είπα, κάθε χώρα μπορεί να αποσύρει ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο από οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση, και έχουμε γι' αυτό το σύστημα των ε, κατόχων κόκκινης κάρτας. Πρόκειται δηλαδή για ένα δικαίωμα ε, κάθε συμμετέχουσας χώρας ε, που εξασφαλίζει και την ανακλητότητα της απόφασης που έχει πάρει για να συμμετάσχει, σε μια επιχείρηση. Εδώ βλέπετε το πορτοφόλιό μας, το χαρτοφυλάκιό μας, διάφοροι στόλοι, έχουμε τακτικούς, στρατηγικούς στόλους, εταιρικούς που μεταφέρουν τα πολύ σημαντικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 160 περιουσιακά στοιχεία τα οποία συγκεντρώνουμε και χρησιμοποιούμε από κοινού και ήθελα να σας πω επίσης ότι ε, η έδρα μας είναι στο Eindhoven όμως έχουμε και 12 αεροπορικές βάσεις ε, αναλογικά ε, είναι κατανεμημένη σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Μία έως τρεις αεροπορικές βάσεις προσφέρει η κάθε χώρα που συμμετέχει στο EATC και εκτελούμε περίπου 60 επιχειρήσεις ε, κάθε μέρα. Εδώ βλέπετε μια διαφάνεια που αποσκοπήσω να σας δείξει ποιο είναι το αποτέλεσμα που αποφέρει η EATC. Εδώ βλέπετε τη συμμετοχή μας και τη συμβολή μας σε επαστολές στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική και στο Αφγανιστάν. Τι κάνουμε, μεταφέρουμε ε, και από και προς τις περιοχές αυτές. Και λέω από και προς διότι η EATC έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο αυτών των ε, περιουσιακών ε, στοιχείων, αλλά επιχειρούμε μόνο από και προς την Ευρώπη. Όταν μιλάμε για αποστολές εντός Μέσης Ανατολής ή εντός Αφρικής, ε, οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλης διοίκησης, όχι τη δική μας. Εδώ βλέπετε τις περιοχές στις οποίες έχουμε εκτελέσει επιχειρήσεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια, 2014 με 2017, 5.000 ήταν αυτές οι αποστολές και κατά τα τέσσερα αυτά χρόνια το 20% των αποστολών αυτό έγινε μέσω ανταλλαγών ατάρες. Αυτό σημαίνει ότι το 20% των αποστολών ωφέλησαν όχι μόνο ένα έθνος, αλλά περισσότερα των δύο. Δηλαδή, περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν ε, σηκώθηκαν μόνο για τη χώρα η οποία τα διέθετε, αλλά ωφελούσαν και ε, σύμμαχες χώρες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διοίκησης Εναέριων Μεταφορών. Και σκοπός μας ε, είναι να αυξηθεί το ποσοστό αυτών των ανταλλαγών ατάρες. Και αφού σας έχω πει λοιπόν τα λειτουργικά, ε, επικεντρωνόμαστε πολύ στην εναρμόνιση, την τυποποίηση και τη διαλειτουργικότητα. Αυτοί είναι οι τρεις τομείς ε, που μας ενδιαφέρουν πολύ και για το σκοπό αυτό ε, εργαζόμαστε στους τομείς της συντήρησης, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. Και γι' αυτόν τον λόγο εκπονούμε μελέτες που έχουν ετηθεί τα κράτη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση και τα οποία ε, και επίσης καταρτίζουμε κανονισμούς, διαδικασίες, διοργανώνουμε εργαστήρια, ομάδες εργασίας, προσφέρουμε κύκλους μαθημάτων σε πανεπιστημιακούς ε, και επίσης διοργανώνουμε και ηλεκτρονικά μαθήματα που απευθύνονται στα, στα 7 έθνη που συμμετέχουν, όχι μόνο όμως σε αυτά, συνεργαζόμαστε και με μη ευρωπαϊκά έθνη. Και η λειτουργική μονάδα ε, αυτή πρέπει να σας πω ότι είναι πλέον το σημαντικότερο περισσοιακό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Διοίκησης Εναέριων Μεταφορών ε, και ε, διαθέτουν ε, την, τα περιουσιακά στοιχεία η Ευρωπαϊκή Διοίκηση σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν ε, συγκεκριμένα εκπονούμε συγκεκριμένα προγράμματα και, και έργα που δραστηριότητες καθοδήγησης ε, που έχουμε καταρτήσει και για το μέλλον. Εδώ προσπαθώ να σας εξηγήσω ποιες, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία μας. Εδώ έχουμε φτιάξει ένα ε, φανταστικό σπίτι, το οποίο αποτελείται από διάφορα τούβλα. Τα κάτω-κάτω τούβλα είναι τα σημαντικότερα διότι αποτελούν το, το θεμέλιο του ίδιου του, του οικοδομήματος που έχουμε ε, φτιάξει. Είναι τα πλέον όρημα και ε, ολοκληρωμένα αν θέλετε και όσο ανεβαίνουμε βεβαίως είναι εξαιρετικά σημαντικά και, και εκείνα τα τούβλα αλλά έχουν ενδεχομένως μια μεγαλύτερη ευελιξία ε, και μια μεγαλύτερη διακύμανση στο κατά πόσο πώς, στο, όσον αφορά το βαθμό στον οποίο ε, χρησιμοποιούνται. Αρχικά λοιπόν αυτό που χρειαζόμασταν ήταν να, να καταρτιστούν ε, συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένα έργα αλλά και να εξασφαλιστεί η βούληση από τα έθνη. Όπως είπα ξεκινήσαμε ως διμερής πρωτοβουλία στην οποία συμμετείχαν στη συνέχεια άλλες δύο χώρες χρειάστηκαν όπως είπα και 10 χρόνια έως ότου καταφέρουμε να καταρτήσουμε και να εκπονήσουμε τέτοιους κανόνες και να ξεκινήσουμε. Επίσης είχαμε το εικονικό νόμισμα, αυτή η μη, η απουσία ροής ε, χρημάτων από τη μία χώρα στην άλλη βοηθά πραγματικά επιχειρησιακά ε, προκειμένου να επιτυχάνονται απτά αποτελέσματα. Γιατί σήμερα όταν τα έθνη ανταλλάσσουν ώρες πτήσης ε, μπορούν να το κάνουν πολύ πιο εύκολα, δεν χρειάζεται να περνούν από μια διαδικασία έγκρισης πραγματικών χρημάτων δηλαδή. Στη δεύτερη σειρά, που είναι επίσης πολύ σημαντική, βλέπετε την ανακλητότητα της, ε, της ε, κάθε μεταφοράς, αλλά και την, τη μεταφορά αξίας και την ανακλητότητα αυτής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι τα ίδια τα έθνη που συμμετέχουν έχουν αποφασίσει να μεταβιβάσουν την εξουσία ε, στην EATC. Κάτι που της δίνει τη δυνατότητα να εκπονεί και να οργανώνει συγκεκριμένες στρατηγικές επιχειρήσεις με το μέγιστο βαθμό αποτελεσματικότητας, αφού της δίνει τη δυνατότητα η κοινή χρήση και η συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων να εξοπλίζει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί δέχτηκαν όμως τα έθνη αυτά να συμμετέχουν και να μεταβιβάσουν εξουσία στην αίτηση. Γιατί, γιατί εξασφαλίζεται η εθνική του κυριαρχία μέσω της ανακλητότητας της διαδικασίας μεταβίβασης εξουσίας. Οποιαδήποτε στιγμή, όπως είπα, μπορεί κάθε χώρα που συμμετέχει να αποσύρει περιουσιακό τη στοιχείο και να ε, χρησιμοποιήσει την κόκκινη κάρτα. Σε οποιαδήποτε στιγμή, λοιπόν, κάθε χώρα που συμμετέχει ε, μπορεί να πει ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να συμμετέχουμε ε, σε αυτή την επιχείρηση. Οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και την τελευταία στιγμή, μπορεί να αποσύρει ε, το, τα στρατεύματά της, το προσωπικό της που συμμετέχει σε μια επιχείρηση, από οποιαδήποτε επιχείρηση. Επίσης, το, η, ATC ενδιαφέρεται και για το μέλλον και μα μας απασχολούν διάφορα θέματα. Τρία έχω επιλέξει για να τονίσω. Θέλουμε να καταστούμε βασικός παράγοντας για την ε, επίτευξη ε, των των, για την επιτυχία των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων και για αυτό το σκοπό είναι απαραίτητο να υπάρξει εναρμόνιση των κανονισμών. Από την αρχή δηλαδή της δημιουργίας της EATC, αυτό ήταν ο βασικός μας, το βασικό μας μέλημα ε, και θα, είναι ένα έργο το οποίο θα συνεχιστεί. Δεύτερο είναι η διπλωματική έγκραση. Ε, της EATC ε, που αποτελεί στόχο προς κατάκτηση ακόμα. Διότι σήμερα, έτσι όπως έχει η κατάσταση, ε, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε πολλά εμπόδια. Θα σας πω κάποιες λεπτομέρειες. Στην, στη διοίκησή μας πολλές φορές λαμβάνουμε ένα αίτημα από μια χώρα που συμμετέχει στη διοίκηση και από εκεί και πέρα ξεκινά η διαδικασία πρέπει να επιλέξουμε καταρχάς τα πλέον κατάλληλα ε, περιουσιακά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Αν λοιπόν η αποστολή είναι να μεταφέρουμε από τη Γερμανία ε, κάτι στην ε, Μέση Ανατολή, χρειάζεται να, κάνουμε, να, περάσουμε, να πετάξουμε πάνω από πολλές χώρες. Και φυσικά για να μπορεί να κάνεις υπερπτήση μιας χώρας χρειάζεσαι διπλωματική έγκριση. Για να τη λάβει κανείς αυτή την έγκριση μπορεί να, να, χρειαστεί, να χρειαστούν δύο μέρες έως τρεις εβδομάδες, ανάλογα με το τι μεταφέρεις και ανάλογα με την ίδια την εκάστοτε χώρα, πάνω από την οποία θέλεις να πετάξεις. Στην αρχή της διαδικασίας βεβαίως γίνεται αυτό, αλλά ε, από τη στιγμή που θα λάβεις αυτήν την ε, διπλωματική έγκριση, αυτή ισχύει για 24 ή 48 ε, ε, ώρες. Αν λοιπόν υπάρξει κάποια βλάβη και δεν καταφέρεις να απογειωθείς, η διπλωματική έγκριση ακυρώνεται. Και εκεί μπορεί να πάρει καινούργια διπλωματική έγκριση ή να αρχίσει να ψάχνει άλλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να σου κάνει την, την μεταφορά στην, στη Μέση ε, Ανατολική. Αυτό είναι πραγματικά μεγάλη δυσκολία. Θα θέλαμε λοιπόν να επιτύχουμε αυτή τη δυνατότητα ε, διπλωματική έγκριση. Κάτι που σήμερα ε, είναι πολύ δύσκολο. Θα θέλαμε λοιπόν να αναγνωριστεί η ATC ω φορέα που μπορεί να λάβει διπλωματική έγκριση, διότι μέχρι στιγμή αυτό που ε, γίνεται είναι ότι κάθε χώρα που συμμετέχει σε μια αποστολή τη σε μια επιχείρηση ATC, είναι υποχρεωμένη η ίδια να λάβει διπλωματική έγκριση. Ε, θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να συστήσουμε ένα γραφείο εδώ στην Ευρώπη ε, και κάθε χώρα με την οποία συνεργαζόμαστε, υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας, σε πάση περιπτώσει, ενδεχομένως και στο πλαίσιο της ΠΕΣΚΟ, να χορηγεί, να χορηγείται σε αυτό το γραφείο η διπλωματική έγκριση. Προφανώς είναι πολύ πιο ε, ισχυρή η θέση μας ε, αν είμαστε αναγνωρισμένοι, ευρωπαϊκή διοίκηση, πολυεθνική και όχι απλά η κάθε χώρα ξεχωριστά μόνη της. Και τέλος, στόχος μας είναι να προωθήσουμε τα πρότυπα και την διαλειτουργικότητα του EATC, κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι η EATC βεβαίως ε, εργάζεται υπέρ των συμφερόντων των 7 εθνών που συμμετέχουν, αλλά και υπέρ ολόκληρης της κοινότητας εναέριων μεταφορών και εναέριου ανεφοδιασμού καυσίνου. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε στη, θέση να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να συμβάλλουμε και να συνδράμουμε ε, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και άλλους ε, συμμάχους και εταίρους όπως είναι η ΕΠΑ. Και όπως είπα ήδη σήμερα Έχουμε καταρτήσει συγκεκριμένα πρότυπα και συγκεκριμένες προδιαγραφές ε, διαλειτουργικότητας, τις οποίες και ε, ανακοινώνουμε και δημοσιεύουμε και ε, κοινοποιούμε και σε άλλες χώρες. Και θα είναι μεγάλη επιτυχία της EATC αν μπορέσουν αυτά τα πρότυπα και οι προδιαγραφές να γίνουν δεκτά και από, άλλους, από άλλες χώρες του πλανήτη. Αυτά. Εδώ σας δίνω μια σύνοψη των δραστηριοτήτων μας για το 2017. Ελπίζω να ανταποκρίθηκα στις προσδοκίες σας, ε, να σας παρουσιάσω και να σας εξηγήσω τον τρόπο λειτουργίας της EATC. Ήταν μεγάλη μου χαρά που ήμουν εδώ και με μεγάλη χαρά επίσης θα δεχτώ τις ερωτήσεις σας και βεβαίως θα απαντήσω και σε αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. for... Ευχαριστώ στρατηγέ για την πλήρη παρουσίασή σας και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους βουλευτές για να συζητήσουμε λιγάκι. Δεν ξέρω αν και ο Γκάλερ θέλει το λόγο ευχαριστώ για τη θαυμάσια παρουσίαση. Χρησιμοποιώ την AATC ε, ως παράδειγμα ενός επιτυχημένου προγράμματος ε, όπου φαίνεται η προσθέμενη αξία της συνεργασίας στον τομέα της ε, ασφάλειας και της άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σύντομα θα θέλατε να μου πείτε ποια είναι η νομική βάση και ποιο είναι το, η βάση συμφωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων. Επίσης, να αναφερθείτε σας παρακαλώ και στην ΠΕΣΚΟ, γιατί έχουμε ακούσει στο Κοινοβούλιο ε, αναφορές ότι η ATC είναι ένας κλασικός φορέας που θα πρέπει να εμπίπτει στην ΠΕΣΚΟ ε, γιατί τότε θα μπορούσαμε να έχουμε και χρηματοδότηση από τον ενωσιακό προπολογισμό. Εγώ θεωρώ ότι αν ξεκινήσουμε έτσι και έχουμε κοινή χρηματοδότηση, είμαι πεπισμένο ότι θα θέλουν και πολύ περισσότεροι να συμμετάσχουν, γιατί ε, αν υπάρχει κοινή χρηματοδότηση, ε, ή μάλλον συγχρηματοδότηση, όλοι αυτοί που από κοινού χρηματοδοτούν, ε, δεν θα είχαν φτάσει στο σημείο που είμαστε και θα ενδιαφερθούν και οι υπόλοιποι. Μήπως λοιπόν θα υπήρχε ενδιαφέρον ε, σε αυτή την περίπτωση να ενταχθούν και άλλοι. Υπάρχουν επίσης ε, παρασκηνιακές συζητήσεις Βλέπω από το χρονοδιάγραμμα που μας δώσατε ότι η τελευταία χώρα που εντάχθηκε εντάχθηκε το 2014. Για ποιο λόγο δεν ε, είχαμε και άλλες επιτυχίες. Η επιτυχία ε, είναι αποδεδειγμένη. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει μεγαλύτερη, ευρύτερη συμμετοχή. Τελευταία ερώτηση για την νομική κατάσταση των ε, στρατιωτών που συμμετέχουν δεν υπήρξαν κάποια προβλήματα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Κάποια οικονομικά προβλήματα με τη συμμετοχή τους. Μήπως έχουν στο μεταξύ επιληθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φρόιν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Δικητά. Ανησυχώ γιατί ο κύριος Γκάλερ σχεδόν μου πήρε τα λόγια από το στόμα, θα, θα την πω την ερώτηση παρόλα αυτά. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ. Αν... Και ξαναδείξτε μου τον τρίτη, τρίτη διαφάνεια με τον ευρωπαϊκό, με το χάρτη της Ευρώπης. Για δείξτε μου λίγο τη διαφάνεια, σας εξηγήσω ποιο είναι το πρόβλημά μου. Ναι, αυτό είναι ο χάρτης της Ευρώπης που θέλω. Αν κοιτάξετε το χάρτη, βλέπετε ότι η Δυτική Ευρώπη είναι εδώ. Δεν υπάρχει ούτε μία χώρα της Ανατολικής Ευρώπης που είναι μέλος στην ATC. Γιατί συμβαίνει αυτό. Κάποιες από αυτές τις χώρες είναι μέλη εδώ και αρκετά χρόνια πια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, να μην σας το εξηγώ περαιτέρω. Κάτι άλλο. Θέλω να αναφερθώ στο τελευταίο σημείο που αναφέρατε. Δηλαδή, όταν ε, κάνεις υπερπτήσεις ε, πάνω από χώρες, χρειάζεσαι μια διπλωματική άδεια. Αν πας ε, στην Μέση Ανατολή, για να πας στη Μέση Ανατολή, περνάς από κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιες τρίτες χώρες. Αλλά υπάρχουν και κοινοτικές χώρες, ενωσιακές χώρες, πάνω στις οποίες γίνονται υπερπτήσεις. Σημαντικό θα ήταν λοιπόν για τι αποστολέ σα για να πετύχετε αυτό το οποίο υπενηχθήκατε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή θα πρέπει να είναι σε θέση να έχει μια κεντρική αδειοδότηση για τέτοιου τύπου αποστολές, ε, δεν θα ήταν καλό να διευθυντήσουμε και αυτά τα θέματα. Συνάδελφοι. Λοιπόν, συνάδελφοι, αν δεν έχετε άλλη ερωτήσεις, να κάνω εγώ. Κύριε ε, στρατηγέ, μιλήσατε για επιχειρήσεις ε, και στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν διατάξεις για αποστολές που ε, προϋποθέτουν, ας πούμε, διαλειτουργικότητα με άλλους εταίρους, ξένους, Αμερικανούς, Καναδούς, Φερρυπίν και άλλους. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου αντιμετωπίστηκαν κίνδυνοι δυσκολίες κτλ. Ποιες ήταν ακριβώς οι δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεράσετε για να γίνουν τέτοιες αποστολές. Δεύτερον, οι ικανότητες που χρησιμοποιούνται. Συνήθως ε, χρησιμοποιείται στόλο κρατικό, πολεμικό, δηλαδή το, το εθνικό πολεμικό ναυτικό ή χρησιμοποιείται ας πούμε και ιδιωτικά σκάφη που ανήκουν σε ιδιώτες πλειοκτήτες. Ανήκουν όλα στο κράτος αυτά τα σκάφη ή όχι. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση για την EMO, για το μνημόνιο ε, συνεννόησης. Ναι, ε, το μνημόνιο συνεννόησης στο οποίο βασιζόμαστε ε, είναι το αρχικό, δεν έχει αλλάξει. Προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με τη συνθήκη. Ακόμα όμως δεν έχουμε φτάσει εκεί. Υπάρχει το αρχικό μνημόνιο. Δεν ξέρω αν θα συμβεί ποτέ να ξεπεράσουμε το μνημόνιο. Δεν ξέρω αν είναι προς το συμφέρον της ε, χώρας νούμερο 1 της Ολλανδίας ή των υπολείπων συμμετεχουσών χωρών. Κάθε χώρα που ανήκει στο EATC χρησιμοποιεί αυτό το μνημόνιο ας πούμε συνεννόησης και η χώρα υποδοχής το δέχεται. Δεύτερο σημείο, το ερώτημα για την ΠΕΣΚΟ, την μόνιμη διαθωμένη συνεργασία. Η δική μας διοίκηση, η ATC, δεν είναι μια ε, ενωσιακή οργάνωση οργανισμός. Είναι η υλοποίηση της θέλησης των ε, ιδρυτικών χωρών, ΨΥΝ, Λουξεμβούργο, Ισπανία και Ιταλία που εντάχθηκαν κατόπιν, Αυτές οι 7 χώρες, 4 είναι 7, ναι μεν είναι μέλη όλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Και εγώ δεν σας λέω ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε αν αποφασίσει ένα κράτος να χρησιμοποιήσει απλώς την ΠΕΣΚΟ. Αλλά εμείς έχουμε και ε, εναέρια μεταφορά και μελέτες και τα λοιπά και ποιος είναι ο λόγος του να συμμετέχεις στην, ΠΕΣΚΟ. Ε, είναι να μεταφέρεις μάχη ομάδες ε, στα πλαίσια μιας επιχείρησης της ΠΕΣΚΟ. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε την ΠΕΣΚΟ, αλλά αυτή τη στιγμή γίνεται μόνο αν το κράτος που αποφασίσει να χρηματοδοτήσει, ας πούμε, ε, ζητήσει από την ATC να το κάνει. Να πει ένα από τα 7 κράτη θα στραφώ προς την ε, η ATC, ή μάλλον προς την ATC, εγώ θα σπονσορά την επιχείρηση ε, εντός της Ευρώπης. Αυτό το έχουμε συζητήσει το θέμα μεταξύ μας. Προσπαθούμε να υπάρξει μία ε, ολοκλήρωση, μία ενσωμάτωση όλων των ευρωπαϊκών χωρών στα πλαίσια της Συμφωνίας Αταρές. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν, έχουμε, δεν είναι εύκολο γιατί δεν υπάρχει και ρευστό στην πραγματικότητα της EADC. Ε, ε, έχουμε αυτό το εικονικό νόμισμα. Είναι μια συμφωνία. Δεν δημιουργούμε τίποτα εμείς. Εμείς λαμβάνουμε ένα αίτημα από ένα από τα 7 κράτη ε, και προβαίνουμε στην υλοποίηση της αποστολής. Χωρίς ρευστό γιατί δεν υπάρχει μια ακόμα χώρα που να έχει ενταχθεί τα τελευταία χρόνια. Κανένα δεν το ζήτησε. Τελευταία χώρα που ζήτησε να ενταχθεί στο EATC ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μας επισκέφθηκαν για πρώτη φορά. Αλλά και μετά το Brexit ε, μας, μας ε, επισκέφθηκε το νούμερο 2 της, του, της ομάδας ε, και εμείς είπαμε ότι θα πρέπει καταρχά να υπάρχει μια πολιτική απόφαση, αλλά θα πρέπει και οι στρατιωτικοί να στείλουν μια επιστολή στην ATC. Γιατί πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε πολιτική απόφαση. Ε, δεν αποφασίζουμε εμεί τίποτα στην ATC. Δεν έχουμε λάβει μια τέτοια επιστολή και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα με τον Brexit. Ε, μπορούν παρόλα αυτά να ενταχθούν, παρόλα αυτά δεν έγινε τίποτα ακόμα Επίσης υπάρχουν και προβλήματα που έχουν οι χώρε. Δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν την ε, σχολή στην ε, Ολλανδία. Προσπαθούμε να βρούμε μια συμφωνία, ούτω ώστε αν είσαι μέλος της ATC να μπορείς να πάρεις άδεια και να θεωρήσεις ότι ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείς να σε κάποιε ε, ακαδημίες, σε κάποιε σχολέ κτλ. Δεν γίνεται όμω. Ε, δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμή. Υπήρχαν προβλήματα για τα μέλη των οικογενειών των στρατιωτών αυτών. Ε, δεν είναι πολλέ οι περιπτώσει με, οι προβληματικές, αλλά προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει με τις οικογένειε των, του προσωπικού, των στρατιωτών δηλαδή. Να πάω τώρα στι ανατολικέ χώρε για να σα απαντήσω σε εσά, κύριε Φραν. Εγώ επισκέφθηκα τις Καναδικές χώρες και υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει μια ιδέα για μια δορυφορική ATC, μια περιφερειακή ATC. Με την Νορβηγία, Φιλανδία, Σουηδία. Ένα σενάριο ένας δορυφόρος εκεί, ένας άλλος στα ανατολικά. Γιατί ποιο είναι το ενδιαφέρον, να είσαι κοντά με τους γειτονέ σου, για να είσαι αποτελεσματικός στις μεταφορές. Γιατί όταν χρησιμοποιούμε στοιχεία περιουσιακά του ατάρες ε, για να κάνουν την αποστολή, ε, καλό είναι ο ένας να μην είναι μακριά από τον άλλον, ε, να μην υπάρχει μεγάλη απόσταση. έχει περάσει χρόνο στην τελευταία αίτηση για ένταξη μια χώρα. Ε, από τη στιγμή που θα το ζητήσει μια χώρα υπάρχει μια περίοδο αξιολόγηση. Σε αυτή την περίοδο θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα υποφεληθούμε και εμένα και, και το κράτο που θέλει να ενταχθεί και εμεί που θα το δεχτούμε. Γιατί θα πρέπει το κράτο να αλλάξει την εσωτερική του οργάνωση, θα πρέπει να αλλάξει τι εσωτερικέ του διαδικασίε και δομέ. θα πρέπει να είναι υποφελέ αυτό για το ίδιο, αλλά και για την ATC. Γι' αυτό τα τελευταία 7 χρόνια δεν αποφασίστηκε να ανοίξει η ATC. Κάποιες ανατολικές χώρες μας επισκέφτηκαν και τους εξηγήσαμε τη διαδικασία, αλλά δεν υποβλήθηκε κανένα επίσημο αίτημα από τις χώρες αυτές για ένταξή τους. Για το δεύτερο ερώτημα, για να ενταχθεί η Αφρική ή η Μέση Ανατολή, ή μάλλον για να πάμε στη Μέση Ανατολή Αφρική θα πρέπει να κάνουμε υπερτήσεις πάνω από ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε αποφασίσει μία διαδικασία για τις υπερπτήσεις. Ε, υπάρχει μία συμφωνία και 15 χώρες έχουν ενταχθεί στην ε, συμφωνία αυτή, έχουν προσυπογράψει. Ναι, 15 χώρες ευρωπαϊκές. Δεν έχουμε πρόβλημα να αυξηθούν οι χώρες, θα ήταν καλό για μας. Εντό τη EATC έχουμε μια πλήρη συμφωνία για όλα τα μέλη τη EATC. Υπάρχει μία μόνο χώρα που δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία αυτή της EATC. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε πρόβλημα με την υπερπτήση πάνω από τη χώρα. Αλλά όταν μπαίνει στην EATC, δέχεσαι με ένα συγκεκριμένο αριθμό ας πούμε άδειας να γίνει υπερπτήση πάνω από την επικρατεία σου. Υπάρχουν κάποια επικίνδυνα αγαθά βέβαια που δεν συνάδουν, που δεν συμμορφούνται με τους κανόνες της ΙΑΤΑ. Εκεί ε, υπάρχει πρόβλημα. Ε, κάναμε όμως μια συμφωνία μεταξύ των έθνων και ως ε, στρατιωτική μονάδα ε, ούτως ή άλλως παραδοσιακά μεταφέρουμε αγαθά που οι εμπορικές ε, αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να μεταφέρουν, άρα το έχουμε ξεπεράσει αυτό το θέμα με τη συμφωνία που έχουμε. Όταν μιλάμε για την υπερπτήση της Σαουδικής Αραβίας ή της Αιγύπτου, ας πούμε, μην ξεχνάτε ότι για να πάρουμε την άδεια υπερπτήσης ε, μπορεί να χρειαστούν τρεις εβδομάδες. Δύσκολο πρόβλημα. Ε, σήμερα διαπραγματευόμαστε κράτος με κράτος. Εάν η Ευρώπη ε, διαπραγματευόταν εκ μέρου 10 ή 15 κρατών, θα ήταν ίσω πολύ πιο χρήσιμο και το διαπραγματευτικό μας χαρτί θα ήταν πολύ πιο καλό. Για να συνεργαστεί τώρα η ATC με τον ΝΑΤΟ. Το ίδιο με αυτό που υπόθηκε για το κράτος, το υπεύθυνο κράτος. Έχουμε κάποιες, κάποια συμφωνία, έχουμε ένα επίπεδο συνένεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, ΝΑΤΟ συνομιλούμε, συνεργαζόμαστε, προετοιμάζουμε την ανάπτυξη των δυνάμεων. αλλά για να γίνει η μεταφορά για το ΝΑΤΟ, για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, θα πρέπει ένα από τα έθνη να ζητήσει αυτή τη μεταφορά που θα πει ναι, εσείς θα μεταφέρετε φορτίο του ΝΑΤΟ. Το πρόβλημα είναι ότι εντός του ΝΑΤΟ κάθε κράτος μεταφέρει τα δικά του στρατεύματα. Για να μεταφέρεις άλλο τύπου πράγματα πρέπει να βρεις άλλους τρόπους. Εγώ πρέπει να μεταφέρω, ας πούμε, τα στρατεύματά μου. Όταν δεν έχω αρκετά τις δυνατότητες να μετά μεταφέρω, τότε ίσως έχει νόημα να στραφώ προς τον Άτομο. Αύριο μεθαύριο, όταν ε, οι αρμοδιότητες μας θα αυξηθούν, μέσα σε 7 ή 10 χρόνια, θα έχουμε πλεονάζον δυναμικό. Και τότε αυτό το πλεονάζον δυναμικό θα μπορούσαμε να το πουλήσουμε στον ΟΗΕ, στον ΝΑΤΟ κτλ. Στο μέλλον μπορούμε να το κάνουμε. Η ATC ε, καλύπτει τα κενά που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο σε αυτά τα 7 κράτη που συμμετέχουν στην ATC. Κάνουμε απλώς πιο αποτελεσματικά τα πράγματα ε, σε επίπεδο η e διαιτησία από ό,τι θα τα κάναν τα 7 αυτά κράτη που συμμετέχουν σε εμά μόνο του. Δεν έχουμε όμω πλεονάζον δυναμικό για να ξεπεράσουμε ας πούμε, την περίμετρο αυτή των 7 κρατών. Δεν έχουμε ας πούμε, δυναμικό να πουλήσουμε. Oh, yes. Yes, your last was about the Η τελευταία ερώτηση αφορούσε τη χρήση των δυνατοτήτων και την ανάθεση σε εξωτερικού φορεί Χρησιμοποιούμε μόνο τον εθνικό στόλο στρατιωτικό ε, στόλο αυτή τη στιγμή με εξαίρεση το Λουξεμβούργο. Σήμερα το Λουξεμβούργο έχει μία σύμβαση με την ε, Luxembourg Airways που είναι μια εθνική εταιρεία για την αεροϊατρική εκένωση. Είναι η μόνη περίπτωση όπου έχουμε αναθέσει σε εξωτερικό φορέα κάτι διότι δεν ανήκουν ε, τα αεροσκάφη αυτά στην αεροπορία του Λουξεμβούργου. Σε όλε τι άλλε περιπτώσει ε, ανήκουν στην εθνική αεροπορία και δεν πραγματοποιούμε outsourcing. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Περιμένουμε ακόμα να ζητήσει κάποιο το λόγο. Να έκανα εγώ, κύριε Στράτη, κάποια άλλη ερώτηση για τις σημερινές συζητήσεις περί στρατιωτικής κινητικότητας ε, για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ΠΕΣΚΟ. Πιστεύετε ότι αυτές οι εξελίξεις θα επεκταθούν ε, ταχαίως ε, με αποτέλεσμα να επεκταθεί ο ρόλος ε, και η εγκαταστάσεις της EATC ή είστε ικανοποιημένοι με το ρόλο όπως έχει προς Και θεωρείτε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει όσο έχει για αρκετό χρόνο. Δεν ξέρω τι να σας πω ακριβώς. Αν με ρωτάει μια από τις χώρες μου, αν μου ζητούσε μια από τις χώρες που έχουμε να συμμετέχω σε μια από τις μελέτες για το έργο στρατιωτικής κινητικότητας στο πλαίσιο της ΠΕΣΚΟ, φυσικά και θα συμμετέχουμε στη μελέτη αυτή. Όπως είπα, και στο πλαίσιο του EUMS ε, ε, υπάρχει αυτό θα προσπαθήσουν είμαι βέβαιος να μας γράψουν σε εμάς σε τέτοια περίπτωση να ε, πραγματοποιήσουν κάποιες συμφωνίες να μας καλέσουν να συμμετέχουμε στις συμφωνίες να λάβουν σωστές συμβουλές από τον EATC αλλά όπως είπα μπορεί να κάνει η EATC ότι δέχονται τα επτα κράτη-μέλη ε, είναι απόφαση δηλαδή των, ε, χρηματο... των κρατών μελών που τη χρηματοδοτούν. Το γνωρίζω αυτό. Ε, τα επτά κράτη αυτά είναι μέλη της ΠΕΣΚΟ, οπότε ναι, απλά εμείς δεν δεσμευόμαστε για κάποια μελέτη. Μπορούμε όμως να δεσμεύσουμε οποιονδήποτε ειδικό μας, αλλά το να εμπλακούμε σε επιχείρηση, αυτό απαιτεί πολιτική βούληση από τα κράτη. Uh, Κύριε Υποστράτη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Σήμερα προσπαθούμε να εστιαστούμε σε μια ε, ποικιλία ε, δράσεων επιχειρήσεων στην Ευρώπη που διεξάγονται τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τα επιμέρους κράτη-μέλη της. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να προβλέψουμε τις αλλαγές, τις μεταβολές στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες ε, για την ε, ενδελεχή σας παρουσίαση, ε, τη λεπτομερή σας παρουσίαση των όλων δράσεων της EATC. Θεωρούμε ότι το εγχείρημα αυτό αποτελεί μια επιτυχία. Ας χειροκροτήσουμε τον υποστράτηγο για τη συμμετοχή του στη συνεδρίασή μας. Το επόμενο σημείο τη ημερήσιας διάταξης για την Κίνα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσει στις 3.30 ακριβώ. Ευχαριστώ.

Colleagues, please be seated. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Thank you. Allow me to restart today's. Uh, ε, ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να συνεχίσουμε με ένα σημαντικό σημείο συζήτηση σε ένα πάνελ ε, που θα, όπου θα συζητήσουμε ε, με την ε, αντίστοιχη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την αντιπροσωπεία για τη σχέση με τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Η Αντιπρόεδρος είναι εδώ ως μέλος της αντιπροσωπείας. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ και το θέμα είναι η προβολή της παγκόσμιας στρατιωτικής ισχύω της Κίνας. Με μεγάλη μου χαρά και τιμή σας παρουσιάζω τρία δικαιοκριμένα μέλη. Ε, πρώτος ο κύριος Κριστόφ Μάνε, αναπληρωτής προϊστάμενος ε, της μονάδας Κίνα, Χονγκ Κόνγκ, Ταϊβάν και Μογγολία. της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Μετά έχουμε την κυρία Εύα Πέισοβα, η οποία έχει ξανάρθει σε συζητήσεις ε, της Επιτροπής ΕΝΤΕ. Φέτος ήδη μας είχε παρουσιάσει την κατάσταση ασφαλείας ε, στην νότια και ανατολική συνική θάλασσα. και σύνοψη και την αποστολή της έδες στην Ιαπωνία. Εστιαστήκαμε σε ζητήματα της περιοχής ε, και σε ζητήματα ασφαλείας εκεί. Όχι μόνο ε, τις κινήσεις του ε, στρατού της Κίνας, αλλά και την τοποθέτηση στρατευμάτων ε, και εξοπλισμό από τη Βορειοκορέα. Η κυρία Εύα Πέισοβα είναι ανώτερη αναλήτρια του EUISS, ε, του Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφαλείας, που έχει εδράσει στο Παρίσι, όπως θα θυμάστε. Και τελευταίος, αλλά ουχή λιγότερο σημαντικός, είναι ο ανώτερος επιστημονικός ερευνητής της RAND Corporation, που έχει έδρα στην Αμερική, ο κύριος Άντρου Σκόμπελ. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στα μέλη του πάνελ και ελπίζω να εποφελθούμε όλοι από αυτή τη συζήτηση. και να γίνει έτσι ένας, και ένας δεύτερος γύρος συζήτησης άμα χρειαστεί. Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Κριστόφ Μανέ. Πάμε κατευθείαν στις παρουσιάσεις. Κύριε Μανέ, έχετε το λόγο. Well, thank you, Mrs. Chair. Thank you for the opportunity. I was given the task to give a general overview before. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Μου ζήτησε θήκη να δώσω μια γενική παρουσίαση πριν περάσουμε στα συγκεκριμένα θέματα ε, και ήθελα να αναφερθώ στην μεταρρύθμιση του λαϊκού απελευθερωτικού στρατού ο πρόεδρος Σιντζιμπίνγκ προχωρά με φιλόδοξα σχέδια για προβολή της κινέζικης δύναμης παγκοσμίω ε, και μέσω της ε, πρωτοβουλίας One Belt One Rule που είναι γνωστή ως ε, BRI της πρωτοβουλίας Μια Ζώνη Ένας Δρόμος θα πρέπει να παρουσιάσουμε τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα ε, στην Κίνα όσον αφορά τις στρατιωτικές της δυνατότητες από το 2015 και μετά. Να αναφέρω δύο πράγματα. Τον Απριλίο του 2015 η Κίνα για πρώτη φορά έστειλε τα στρατεύματά της στο εξωτερικό στην Ιεμένη, μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, ώστε να εκενώσει τους δικούς της πολίτες. Το 2015 η Κίνα διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία για πρώτη υπεράκτια, ε, υπερπόντια στρατιωτική βάση στο Τζιμπουτί για τα κινέζικα πλοία που ξεκίνησε τις δραστηριότητες της ε, πέρυσι. Όλο ένα ακούμε φήμες και για άλλες βάσεις, για άλλες διαπραγματεύσεις που αφορούν πιθανώς μια βάση στην Αμίμπια, μια άλλη στο Πακιστάν, στο Κοντάρ και άλλη μια στη Σρι Λάνκα. Το Δεκεμβρίο του 2015 το Εθνικό Λαϊκό ε, Συνεδρίο της Κίνας πέρασε ένα νόμο που ε, νομιμοποιεί τις αντιτρομοκρατικές δράσεις στο εξωτερικό και στα τέλη του 2015 η Κίνα ξεκίνησε μια άνευ προηγουμένου ριζική στρατιωτική μεταρρύθμιση με σκοπό την περαιτέρω αύξηση του ρόλου του ναυτικού μειώνοντας ε, την αναλογία των επίγειων στρατευμάτων, παρέχοντας τη δυνατότητα ε, διεξαγωγή ε, τεχνικού πολέμου επίπεδου του 21ου αιώνα ε, με την καθιέρωση συνδυασμένων διοικήσεων για δράσεις από διαφορετικά κομμάτια του στρατού όπως στη Δύση. Αντικαθιστώντας δηλαδή το παλιότερο σύστημα περιφερειακών διοικήσεων. Το 2017 είχαμε τη δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης που εστιάστηκε στο να γίνει το PLA πιο ευέλικτο ε, μειώθηκε μειώθηκαν ε, οι στρατιωτικές ομάδες από 18 σε 13 ε, και επεκτάθηκαν οι νέες και οι κινητές δυνάμεις μάχης όπως για παράδειγμα ελικόπτερα και ναυτικές δυνάμεις για άλλη μια φορά η μεταρρύθμιση επέδρου στο PLA να διεξάγει πιο αποτελεσματικέ δράσει στο εξωτερικό αντί απλά να υπερασπίζεται την ε, ε, Κίνα. Επίση, ε, εξυγχρονίστηκε η στρατιωτική εκπαίδευση. Βάσει πιο ρεαλιστικών προσδοκιών, τον Σεπτέμβριο του 2017 η Κίνα ολοκλήρωσε την στρατολόγηση επιπλέον 8.000 ειρηνευτικών δυνάμεων των ΗΠΑ, δίνοντας ε, σε, στις ομάδες της τη δυνατότητα να αποκτήσουν πραγματική εμπειρία μάχης. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η Κίνα ε, απορρίπτει την ιδέα της παγκόσμιας ηγεμονίας και δεν δύναται. Θεωρούμε δηλαδή ότι δεν πρόκειται να δοκιμάσει το στρατιωτικό το στρατό της, αλλά απλά το διατηρεί ε, για επίδειξη ισχύω, όπω συμβαίνει στην αντιπαράθεση με την Ινδία. Τη λείπει η εμπειρογνωμοσύνη να διεξάγει πολέμου, μπλέκεται σε ειρηνευτικέ διαδικασίε, ε, σε ειρηνευτικέ επιχειρήσει, όπω είπα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, που μοναδικό ε, απότερο στόχο έχει την επιβίωσή του, δεν θα μπορούσε να αντέξει μια αποτυχημένη στρατιωτική επιχείρηση. Θα φαινόταν ως αδυναμία, θα μείωνε την λαϊκή υποστήριξη της προβολής Κίνας στο εξωτερικό, και θα υπονόμευε τη φήμη του, τη φήμη της Κίνας ως παγκόσμιας δύναμης. Το κογκρέσο του κόμματος τελευταίο ε, ε, έδειξε ποιοι είναι οι στόχοι, ανέφερε τους στόχους της Κίνας ε, υπό τον Σιν Τζιμπίνγκ ταυτόχρονα ο στρατός ορίστηκε ως ο στρατός του κόμματος το λέει είναι ο στρατός του κόμματος ουσιαστικά του κομμουνιστικού κόμματος Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός. Όλα αυτά στον δρόμο για την οικοδόμηση μιας πλέον σοσιαλιστικής ε, Κίνας. Ο στόχος που είναι η πλήρης μηχανοποίηση ε, μέχρι το 2020, η πλήρης εξυγχρονισμός μέχρι το 2025 και παγκόσμιου επίπεδου δυνάμεις μέχρι το 2050 συντονίζεται περίπου με την ιδέα του η Κίνα να γίνει μια μεγάλη σύγχρονη σοσιαλιστική χώρα. Ο στόχος αυτός φυσικά είναι μακροπρόθεσμος με τις προσπάθειες και τις φιλοδοξίες της Κίνας ε, να εξελιχθεί μαζί με ε, την ε, μετατροπή του λαϊκού απελευθερωτικού στρατού. Όλα αυτά μαζί με μια πιο αποφασιστική εξωτερική πολιτική συμπεριλαμβανομένου του στόχου να ε, εξαλειφθούν οι προσπάθειε για την ανεξαρτησία τη Ταϊβάν. Ωστόσο, η, Κίνα δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτικέ δυνάμει στην εξωτερική τη πολιτική, αλλά χρειάζεται τι δυνατότητε για να την διασφαλίσει. Χρειάζεται, όπω είπα, ε, κάποιου οικονομικού στόχου, όπως αναφέρονται στις σχετικές φιλοδοξίες. Και τώρα ε, και τώρα θα περάσω στις ε, επίκες διαδρομές που χρησιμοποιούνται για την προβολή του λαϊκού απελευθερωτικού στρατού. Όπως αναφέρθηκε η Κίνα, δεν έχει την ε, ε, στρατιωτική δύναμη που απαιτείται και έτσι ο λαϊκός απελευθερωτικός στρατός δεν μπορεί να αναπτυχθεί δίπλα σε παρόμοιες στρατικές δυνάμεις όπως στη Ρωσία, στην Ασία. ή να σταθεί στο ύψος της ε, περίπλοκης ισορροπίας δυνάμεων ε, στην Ασία με Ινδία, Αφγανιστάν κτλ. Παρότι ξεχωρίζει σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ιστορικά η Κίνα υποστηρίζει το δόγμα της περιπλοκης ισορροπια δυναμεων στην ασια με ινδια διαφορίας. εξωτερικη πολιτικη ιστορικα η κινα υποστηριζει το δογμα τη μια διαφορία. αλλα καθως της μη επέμβαση χρησιμοποιεί και άλλα μέσα Και θα σας δείξω τώρα τι εννοώ. Το Uber είναι ουσιαστικά έχει, είναι πολύπλευρο. Είναι μια επιτυχής δημόσια εκστρατεία που υποστηρίζει όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες στο εξωτερικό. Ουσιαστικά αλλάζει το χαρακτηρισμό μιας προϋπάρχουσας υποδομής. Αποτελεί και ένα ε, έργο οικονομικής ολοκλήρωσης ε, με την Κίνα στο κέντρο της. Δημιουργήθηκε προϊθανότητα για εσωτερικές αιτίε. Από οικονομική άποψη είναι ένας τρόπος εξαγωγής ε, το υπερβολικού, της περισσίας δυναμικού της Κίνας. Γεωστρατηγικά χρησιμεύει επίσης και ως τρόπος ε, ένταξη των δυτικών περιοχών της ε, Κίνας όπω το Σιντζιάν ε, που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα που είναι οικονομικά πιο πίσω από την υπόλοιπη Κίνα αλλά που αντιστοιχούν στο, σε πάνω από το 1 πέμπτο της παραγωγής κάρβουνου και φυσικού αερίου και πετρελαίου της Κίνας. Το Σιντζιάν είναι επίσης μια αναπόφευκτη επίγεια οδός προς την υπόλοιπη και την Ευρώπη. Στη Δύση οι γειτονικέ χώρε της Κίνας ε, ε, πολιτισμικά είναι ε, κοντινέ στο Σιντζιάνγκ. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτός ο στόχος εξουδετερώ πιθανών ασφαλών λιμένων. Ο στόχος είναι επίση. είναι η επέκταση προς δυσμάς ώστε να αποφευχθεί ο περιορισμός των αποθαλάσσιες ε, περιοχών, των παραθαλάσσιων περιοχών ε, από ε, μέχρι την Ινδία ώστε να ανοίξει ο διαδρόμος προς το Πακιστάν επίσης και αυτός είναι ένας τρόπος ώστε η Κίνα να διαφύγει το δίλημα των στενών της Μάλακα. Τέλος υπάρχει και η ψηφιακή διάσταση και ο συνδυασμός ε, των, ε, της προβολής δυνάμεων. Η Κίνα πουλά ταυτόχρονα ε, τεχνολογία πληροφοριών σε κινέζικα κράτη, ενώ ταυτόχρονα εξάγει ένα δόγμα ψηφιακής κυριαρχίας, κυριαρχίας του κυβερνοχώρου που πολλά κράτη-μέλη θέλουν να υιοθετήσουν. Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις αντί για τον πόλεμο, η Κίνα βρίσκει και άλλους τρόπους να προβληθεί ως παγκόσμια δύναμη. Αναφέρα την αντιτρομοκρατία ε, με την άδεια που δόθηκε το 2015 σε θέματα αντιμετώπισης τη τρομοκρατίας από το δεκαετία του 1990 προτεραιότητα για τις ε, υπηρεσίες ασφαλείας της Κίνας ήταν η διμερή συνεργασία της Κίνας με τα κράτη της ευρύτερης Κεντρικής Ασίας εγκύτητα με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και ισχυρή συνεργασία με το Πακιστάν. Στις αρχές του 2016 η Κίνα, το Τατζικιστάν, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν δημιούργησαν ένα τετραμερή μηχανισμό συνεργασίας ε, για από καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι πωλήσει όπλων επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο. Στις αρχές του 2015 η Κίνα παρήχε στο Τουρκμενιστάν και δεχομένως στο Ουσμπικιστάν εξελιγμένης τεχνολογίας ε, συστήματα αεράμενας που ε, αποτελούν τη μεγαλύτερη ε, συμφωνία όπλων που είχε στην Κεντρική Ασία μέχρι στιγμή η Κίνα. Το Πακιστάν φυσικά είναι ο σημαντικότερο πελάτη κινέζικων όπλων. Αντιστοιχεί στο 1 τρίτο των πουλήσεων όπλων τη Κίνα από το 2013 μέχρι το 2016. Εδώ, ωστόσο, ο ανταγωνισμός με τη Ρωσία περιορίζει την πίστη της Κίνας. Ε, φαίνεται από την περίπτωση του Τατζικιστάν. Μετά από τις πωλήσει ε, στρατιωτικών όπλων στο Τατζικιστάν το 2014, ε, αξίες πολλών εκατομμυρίων, η Ρωσία υποσχέθηκε στο Τατζικιστάν τεράστια ποσότητα μαχητικών αεροσκαφών το 2016. Συμπερασματικά η Κίνα συνεχίζει να επιδιώκει μια σχετικά παθητική ξένη πολιτική. Η κινέζικη πολιτική και διπλωματία παραμένει επικεντρωμένη στον εαυτό της και η συμμετοχή στην παγκόσμια διακυβέρνηση είναι ελάχιστη και διατηρείται τακτική χωρίς καμία στρατηγική. Η κινέζικη διπλωματία ουσιαστικά το μόνο που την απασχολεί είναι οι επιχειρήσεις. Αν εξετάσει κανείς ε, τη σύνθεση των αντιπροσωπιών της Κίνας ή του Πρωθυπουργού του Εξωτερικού, του Πρόεδρου του Εξωτερικού, ε, αποτελούνται συνήθως από επιχειρηματίες, πρόεδρους επιχειρήσεων σε θέματα ε, ενέργειας, ε, συζητούν θέματα εμπορικά και επενδυτικά. Αυτή η του πρωθυπουργου του εξωτερικου του προεδρου στο εξωτερικό αποτελουνται συνηθως απο επιχειρηματιες προεδρους επιχειρησεων σε θεματα ε ενεργειας διπλωματία δεν ε, χαίρει διεθνούς ε, ε, σεβασμού και αρχίζει να δημιουργεί όλο και περισσότερο ε, κριτική παγκοσμίω, ειδικότερα στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική. Μακροπρόθεσμα όμως φαίνεται ότι η επίσημη μη παρεμβατική πολιτική της Κίνας θα αλλάξει. Η Κίνα αρχίζει να ευθυγραμμίζει τις στρατιωτικές της δυνατότητες με την κλίμακα της οικονομίας, της επικράτειας και του πληθυσμού της. Και έχει επιτύχει εντυπωσιακή πρόοδο ενισχύοντας τη δυνατότητά της να προβάλλει στρατιωτική δύναμη σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή είναι μια φυσική αναπόφευκτη διαδικασία, ε, παρότι έχει καθυστερήσει και σχετίζεται στενά με τους μακροχρόνιους στόχους του Κομμουνιστικού Κόμματος να καταλήξει σε κατάσταση ε, Παγκόσμια δύναμη. Στο μεταξύ χρησιμοποιεί δυνάμεις όπως το ΟΜΠΕΡ και άλλες επιχειρήσεις ε, μη πολεμικέ, μη στρατιωτικέ για να προβάλλει τη δύναμή τη. Ευχαριστώ. Thank you, sir. Ευχαριστώ. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Εύα Πέισουβα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, την εισαγωγή σας, την πρόσκληση για να μιλήσω για αυτό το ενδιαφέρον θέμα σε ένα τόσο ενδιαφέρον ακροατήριο. Όπως και άλλοι ομιλητές, μου ζητήθηκε να μιλήσω για την, για την προβολή της ε, κινέζικης θαλάσσιας δύναμης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, μου ζητήθηκε να μιλήσω για τη θαλάσσια δύναμη, γιατί έχω τέτοιο background, αλλά γιατί η θαλάσσια ο θαλάσσιος βραχίωνας έχει μεγαλύτερη παγκόσμια εμβέλεια και τον αισθανόμαστε περισσότερο εδώ στην Ευρώπη. Δεν είναι δύσκολο έργο αυτό. περάσω στο ψητό. Ίσως θα υπάρξουν κάποιες επικαλύψεις με τα όσα ακούσατε προηγουμένως. Θα σας πω ποιες είναι οι τελευταίες και να σας δώσω και κάποιες κλίδες ανάλυσης της θαλάσσιας ισχύω της Κίνας και της επιπτώσεις στην ασφάλεια για την Ευρώπη. Ο κ. Μανέ αναφέρθηκε στο, στη μεταρρύθμιση του Κινέζικου στρατού το 2014. Θεωρούμε ότι είναι ορόσημο και βασική κίνηση στην στρατιωτική πορεία της Κίνας, γιατί εστιάζει περισσότερο στα ποιοτικά στοιχεία το στρατιωτικών της δυνάμεων. Ε, έγινε με μεγάλη αναδιάρθρωση των ενόπλων δυνάμεων. Ε, διορέθηκε η κεντρική διοίκηση σε 15 υποδιοίκησεις. Ε, Υπάρχει λιγότερο μονοπόλιο και μεγαλύτερη διαφάνεια στην διοικητική αλυσίδα. Ε, οι τρεις βραχίονες του στρατού ε, που είναι ε, οι χερσαίε δυνάμεις, οι εναέριες δυνάμεις και οι θαλάσσιες δυνάμεις εμπλουτίστηκαν άλλε δύο. Μία που ασχολείται με την κυβερνοάμυνα και η άλλη με τον εναέριο χώρο. Μιλάμε για ένα άρδιν εξυγχρονισμό των κινέζικων στρατιωτικών δυνάμεων ε, και πρέπει να σας πω ότι δεν έχουν κάτι τέτοιο όλοι οι στρατοί σε τον κόσμο. Ε, ε, δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι υπόδειγμα, αλλά σίγουρα είναι ενδιαφέρον ως μοντέλο. Ως τμήμα του εξυγχρονισμού αυτού βλέπουμε ότι υπάρχουν μειώσεις του προϋπολογισμού και του προσωπικού αποφάσισε να κόψει ε, με έως 2 εκατομμύρια άτομα. Ε, μιλάμε για διοικητικό προσωπικό ε, και για να μειώσει το διοικητικό άφθος. Δεν ε, μείωσε τις μάχημες ε, μονάδες. αποφάσισε να βελτιώσει την ευημερία των στατευμάτων με βελτίωση των, του μισθού, αύξηση του μισθού κατά 20% ή μέχρι 20% και δυνατότητες μετά να μεταπηδήσουν σε άλλες κρατικές επιχειρήσεις αφού φύγουν από το στρατό. οι κριτικές που ασκήθηκαν στην Κίνα ήταν ότι ήταν παλιωμοδίτικο ο στρατό, ε, έμοιαζε με τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό ο στρατό γίνεται πολύ πιο μοντέρνο, με μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία. Προπολογισμό. Ο προπολογισμό συχνά είναι το πρώτο πράγμα που εξετάζουμε όταν αναλύουμε το, τη στρατιωτική ικανότητα και την ισχύ μια χώρας και συχνά είναι το απότατο παράδειγμα ε, οικοδόμησης ε, ισχύω της Κίνας ε, συγκριτικά η τάση αυτή υπάρχει εδώ και 20 χρόνια, αλλά σε σχέση με το 2015 υπάρχει μια μικρή επιβράδυνση από αύξηση σε διπλό ψηφίο πάνω από 10%. Έχουμε τώρα ε, από το 15 και μετά 7%. 7% ε, αύξηση δεν είναι λίγο, δεδομένης της κινέζικης οικονομίας, του μεγέθους. Μιλάμε για 40 δισεκατομμύρια ευρώ αύξηση. Ε, στην γραφική παράσταση εδώ βλέπετε τις α, διαφορές. Ε, μιλάμε για τα επίσημα στοιχεία εδώ. Μπορεί να φτάσουμε και στα 270 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος. Αύξηση μιλάμε. Αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα που δαπανά για, τις, για την αμυνές μετά τις Ηνωμένε Πολιτείες. Οι Ηνωμένε Πολιτείες θα πούν 36%. Ε, τρίτη θέση, στην τρίτη θέση Αουδική Αραβία. Ο προπολογισμό ξοδεύεται, ε, γίνεται ισοκατανομία του δαπανών του προπολογισμού ανάμεσα στους διάφορους τομείς ε, χερσαίες δυνάμεις, αναέρειες δυνάμεις και θαλάσσιες δυνάμεις. Το, ο στόλος και η αεροπορία είναι οι δύο βραχίονες του στρατού που λιγάκι έχουν κάποια προνόμια. Να μιλήσω για το ποιοτικό στοιχείο. Τώρα μπαίνουμε στις λεπτομέρειες, ε, στο... οι Κινέζοι μπαίνουν στις λεπτομέρειες στο σχεδιασμό. Ε, εδώ βλέπετε τα γυμνάσια του Κινέζικου Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού. Το 16 βλέπετε μια έκρηξη ε, γυμνασίων, κατάρτισης, ασκήσεων ε, όπου συμμετέχουν και συνεργάζονται ξένες αθλητικές δυνάμεις, κυρίως ασιατικές. Η Νοτιοανατολική Ασία, μάλιστα, είναι ο πρώτος εταίρος και η Ευρώπη είναι στην δεύτερη θέση ε, στη συμμετοχή σε στρατιωτικά γυμνάσια. Δεν μιλάμε μόνο για κατάρτιση, μιλάμε για επισκέψεις επίσης ανώτατων αξιωματούχων, στρατιωτικών αξιωματούχων πάλι. Πολύ μπροστά σε σχέση με τους Αμερικάνους είμαστε σε συνεργασία αυτή ή τους Ρώσους. Λοιπόν, γιατί τα κάνει όλα αυτά η Κίνα. Τώρα ας περάσω καταρχάς ε, στον αμυγός θαλάσσιο τομέα. Ε, γίνεται μια διάκριση των θαλασσών στις ε, θάλασσες που είναι κοντά και στις μακρινές θάλασσες. Είναι σαφέστερη η διάκριση αυτή. Η εθνική ασφάλεια και Παρατοσιακές αμυντικέ ε, συνιστώσει είναι προφανείς. Πιστεύει η Κίνα ότι οι βασικέ απειλέ έρχονται από το εξωτερικό και όλη η πραγματική ισχύς ε, και το στρατιωτικό δυναμικό ε, σχεδιάζεται για να υπερασπιστεί η Κίνα το, την αθρική της αρτεραιότητα και την, σε περίπτωση μείζωνος επίθεσης. Και η μάχη για την Ταϊβάν αναφέρεται συχνά ε, στο θαλάσσιο αμυντικό δόγμα, προφανές είναι αυτό, ε, κυριαρχικά συμφέροντα και δαφική ακαιρεότητα στην ε, θάλασσα της Κίνας και στην γειτονία της είναι πυρηνικά θέματα, αδιαμφισβήτητα και θα θέλουν να υπερασπιστούν όλα αυτά τα εδάφη και φυσικά οικονομική εκμετάλλευση. Αυτή είναι τα, αυτά είναι τα συμφέροντα στις γειτονικέ θάλασσες και τα εξασφαλίζει όχι μόνο το ναυτικό, αλλά οι 7 δράκοντες που έχει η Κίνα, όχι μόνο το ναυτικό, αλλά η υπηρεσία για την θαλάσσια για την πολιτική θαλάσσια εφαρμογή, διάφορες πολιτοφυλακές και διάφοροι άλλοι οργανισμοί και φορείς. Αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να κοιτάξουμε τώρα και, την, τα παγκόσμια εργαλεία και κίνητρα ε, της Κίνας θέλει καταρχάς να προασπιστεί το εμπόριό της, τις γραμμές επικοινωνίας μέσω των οποίων διεξάγει αυτό το εμπόριο. Λογικό, η Κίνα εξαρτάται από το διεθνές εμπόριο. Ε, είναι παγκόσμια δύναμη, εισάγει το 90% της ενέργειάς της από τα, τους θερματικούς σταθμούς στην Μέση Ανατολή και εξάγει όλα της τα βιομηχανικά αγαθά. Με την πρωτοβουλία αυτή, ε, μία ζώνη, ένας δρόμος, ε, θέλει να προστατεύσει και την ε, κινέζικη διασπορά και να πετύχει το καθεστώς της παγκόσμιας δύναμης. Προφανώς. Όταν κοιτάξουμε ε, τις ικανότητες που έχει στις μακρινές θάλασσες, τα μπλε ύδατα όπως λέγονται, εγώ δεν ξέρω αν συμφωνώ 100%. Δεν διαφωνώ βέβαια 100% με του συναδέλφου που λένε ότι η Κίνα δεν έχει την ε, σκληρή δύναμη για να τα όλα αυτά. Γιατί με βάση τις προβλέψεις για το 2020 η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη θαλάσσια δύναμη στις μακρινές θάλασσες παγκόσμια. Είναι αυτά εδώ κάποια παραδειγματάκια που βλέπετε για να βλέπετε, να δείτε, ε, βλέπετε πόσους πόσα μεταγωγικά ε, ελικοπτεροφόρα και αεροπλανοφόρα ε, φτιάχνει η Κίνα. Έχει, έχει αντιτορπιλικά ε, αντίστοιχα με τον Αμερικανών, απόλυτα συγκρίσιμα, έχει... Ε, υποβρύχια με πυρηνική ισχύ Βλέπετε εδώ ότι εμείς και το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί πόρο απέχουμε. Η Ιαπωνία έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν έχει αεροπλανοφόρα μεταγωγικά. Έχει μόνο ελικόπτεροφόρα που έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν αντίστοιχου στόχου. <laughs> Έχουμε κάνει δικές συνεδριάσεις ε, που ασχολούνται με τη θαλάσσια γειτονία της Κίνας, ε, η θάλασσα της Ανατολικής Κίνας και της Νότιας Κίνας είναι γειτονικές θάλασσες, να το πω έτσι απλοϊκά, έτσι. Για να σας προσανατολίσω. Δεν χρειάζεται να μπω σε πολλές λεπτομέρειε γιατί η θάλασσα τη Ανατολική Κίνα. Ε, πρόκειται για μια διμερή διαμάχη που έχει η Κίνα με την Ιαπωνία, όπου μπλέκονται θέματα ε, συνόρων και κυριαρχίας είναι ε, αλληλοσυνδεδεμένα αλλά και διακριτά αυτά τα θέματα και είναι καυτό θέμα. Ε, μήλο, του, μήλο της έριδος τα τελευταία χρόνια. Ε, υπάρχει ένταση και κλιμάκωση από το 12 με ε, δήλωση που έγινε το 2013 και εντοπισμό της, των ζωνών που είναι κινέζικα κτλ. Ε, αν πάτε στην Κίνα, ε, θα δείτε ότι κάποια κέντρα κατάρτισης και εκπαίδευσης του ναυτικού ε, χρησιμοποιούν για την κατάρτισή του τους ε, μοντέλα για το πώς θα ανακτήσουν εδάφη, φερρυπίν, τέτοιου τύπου εδάφη. Η θάλασσα της Νότιας Κίνας φυσικά είναι πολύ πιο αμφισβητούμενο περίπλοκο παράδειγμα με αλληλεπικαλύψεις. Πολλοί διεκδικούν κυριαρχία, έξι χώρες, έως έξι χώρες διεκδικούν και δικαιώματα εκεί. Είχαμε μια ειδική σύνοδο που κάναμε γι' αυτό και δεν θα μπω σε λεπτομέρειε για αυτή τη θάλασσα, ε, γιατί μιλήσαμε για το θέμα αυτό πριν από ένα χρόνο. Έκτοτε δεν έχουν βελτιωθεί πολύ τα πράγματα. Έχουν υπάρξει βελτιώσει μεταξύ τη ΑΖΕΑΝ και τη Κίνα για τον κώδικα διοντολογία, αλλά στο μεταξύ η, η ανάπτυξη δυνάμεων στα νησιά και η στατιωτικοποίηση συνεχίζεται, δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό που είναι σημαντικό στην θάλασσα της Νότιας Κίνας είναι ότι μας δείχνει πώς συμπεριφέρονται οι Κινέζοι στην πραγματικότητα. Μας δείχνει μια κλίδα ανάγνωσης. Είναι παράδειγμα και μας δείχνει πώς πάει τους κανόνες, πώς τους παραβιάζει, πώς εκφοβίζει τους υπόλοιπους, τις μεθόδους εκφοβισμού που χρησιμοποιεί τα φάσματα τα οποία χρησιμοποιεί στο αφήγημά της κτλ. Και, και ε, φωτίζει και τα όσα κάνει και ένα αλλού. Ε, αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον ίσως για μας, για τη σημερινή μας συνεδρίαση, είναι τι γίνεται όταν περνάμε πιο κοντά στις δικές μας περιοχές, πιο δυτικά δηλαδή, ε, στην περιοχή Ινδίας Ειρηνικού, που ήταν σε επιχαίους τίτλους πρόσφατα. Και έχουμε μια ε, δαθμία ανάπτυξη δυνάμεων στον ειδικό ωκεανό. Ξεκίνησε το 2008 αυτή η ανάπτυξη. Ε, επιχειρήσεις ε, κατά τη πειρατεία, ε, όπου στην πραγματικότητα η Κίνα υπεράσπιζε τι δικέ της ναυτικέ οδούς, λογικό και δικαιολογημένο. Σιγά σιγά όμως ε, βοηθούσε ας πούμε, τις χώρες περιοχής για να απτύξουν τι ε, του υποδομέ υποδομές, που στην αρχή ε, αναφέρανε τη στρατηγική αυτή ως ε, το, το κομπολόι από, τις, ε, από τα μαργαριτάρια. Σρι Λάνκα, Μιανμάρ, Μπαγκλαντές, Πακιστάν. Και σιγά σιγά Ανατολική Αφρική. Ανάπτυξη δηλαδή λιμένο σε αυτές τις όλες τις περιοχές που σας ανέφερα. Στο μεταξύ, αυτή η τάση γίνεται όλο και πιο ανησυχητική. Φυσικά εξαρτάται το, την οπτική γωνία του καθενός. Αλλά για την Ινδία σίγουρα είναι προβληματικό αυτό. Ε, πολέμηση τη πειρατεία. Πολύ ωραίο. Καλό και άγιο. Αλλά έχουν περάσει 10 χρόνια. Η Κίνα έχει συνοδεύσει πάνω από 6.000 πλοία ε, και έχουν υπάρξει χιλιάδες επιθέσεις ε, ε, χίλιες, δύο χιλιάδες κτλ. Και αυτή είναι μια τέλεια ευκαιρία ε, για να υπάρξει εμπλοκή της Κίνας ε, σε διεθνές επίπεδο ε, έτσι. Πολύ ωραία. Για να καταπολεμηθεί η πειρατεία. Αυτό είναι καλό και άγιο. Αυτό που δεν είναι τόσο καλό και τόσο άγιο είναι ότι χρησιμοποιούν αμάχους ή υποδομές μη στρατιωτικέ για στρατιωτικού σκοπού. Είχαμε επισκέψει, α πούμε, ε, υποβρυχίων στη Σιλάνκα και στο Πακιστάν, που κάποιες από τις περιφερειακές δυνάμεις θεωρούσαν ύποπτα. Εφτά τέτοιε επισκέψει έγιναν. Από αυτέ που ξέρουμε, έτσι. Που, εφτά που ομολόγησαν οι Κινέζοι. Ε, υπάρχει η ναυτική βάση στο Τζιμπουτί, το 2017 και το 2016 που λέει η διαφάνεια. Εν συνεχεία, επίσημα υποτίθεται θα υπήρχε επιμελητία, επιμελητική υποστήριξη. Και μόλι τον, Νοέμβριο 2017 έγινε γυμνάσια με πραγματικές σφαίρες, πραγματικά πυρά. Τι δουλειά έχουν τα πραγματικά πυρά στην επιμελητία. Ε, στον ε, Δυτικό Ινδικό Ωκεανό έγιναν ασκήσει. Και κατά τύχη τον Αύγουστο μία άγνωστη χώρα στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό συμμετείχε. Είχαμε τότε την ε, κλιμάκωση της σύγκρουσης ε, για το Όκλαμ με την Ινδία. Υπήρχαν και διάφορες δραστηριότητες, όλο και περισσότερες, ε, περιπολίες στον Ινδικό Ωκεανό. Είναι τμήμα και αυτά της εξίσωσης. Κινέζικα γυμνάσια στη Μεσόγειο τον Ιούλιο του 2007 μέχρι και τη Βαλτική για να ε, συμμετάσχει σε γυμνάσια των Ρώσων η Κίνα. Αυτά τα είδαμε και θα πρέπει να τα συνηθίσουμε μάλλον. Θα γίνουν όλο και πιο συνήθι και μπανάλ και κλασικά από εδώ και πέρα. Και τώρα θα πάω στο, στο δόγμα μία ζώνη, ένας δρόμος. Αλλά πρέπει να σας πω από την ε, θαλάσσια σκοπιά είναι ένα γεωπολιτικό project μεγάλης εμβέλειας. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι είναι ελκυστικό σχεδόν για όλους. Όταν ε, μιλάμε στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας υπάρχει ενθουσιασμός για αυτό το πράγμα. Αλλά, συγγνώμη, κανένας δεν είναι ενθουσιώδης, αλλά κανένας τον στην Νότιο-Ανατολική Ασία ε, θεωρούν ότι είναι δεδομένο η άνοδος της Κίνας. Ε, θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, να χρησιμοποιήσουν έτσι αυτή την τάση ας πούμε και ίσως να υποφεληθούν λιγάκι από αυτή την ευημερία που γεννιέται. Οι μικρότερες χώρες στην ε, Νότια Ασία ε, χρησιμοποιούν την Κίνα για να αντισταθμίσει τη δύναμη της Ινδίας. Ε, και έχουν παραδοσιακά μία θετική εικόνα για την Κίνα. Ε, Μέχρι και την Ευρώπη φτάνει αυτή η θετική εικόνα. Βλέπετε τι έγινε στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες όπου κάποιες επενδύσεις σε έργα υποδομών που έκαναν οι Κινέζοι αφορούν πια αυτές τις χώρες, στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, αυτό που είναι ενδιαφέρον και ίσως είναι η πιο σημαντική διαφάνεια από αυτές που σας παρουσιάζω είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την στρατιωτική όταν μιλάμε για προβολή στρατιωτική ισχύω, εγώ τη λέω υβριδική, ε, το κάνω για λόγου ευκολίας και τεμπελιάς. Πρόκειται για συνδυασμό στην πραγματικότητα οικονομικής, διπλωματικής, πίεσης, μαζί με στρατιωτική ισχύ και πίεση. Ε, μόνο αν κοιτάξετε το στρατιωτικό σκέλος ε, δεν θα καταλάβετε πλήρω την εικόνα. Δεν είναι συμβατικές οι μέθοδοι. Ε, μιλάμε για μεθόδους, ε, τη μέθοδο του σαλαμιού, ας πούμε, του κατακαιρματισμού που χρησιμοποιούμε στην Κινέζικη θάλασσα, θάλασσα τη Νότια δηλαδή. Δεν θα τα ξαναπώ αυτά. Αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό είναι ότι με τις διμερείς διαπραγματεύσεις που κάνουν με μικρότερες χώρες, Μπαίνουμε σε σχέσεις εντελώς ασύμετρες, βαθιά ασύμετρες. Και δεν θα έλεγα ότι είναι επιθετικές, αλλά στην πραγματικότητα οι Κινέζοι ε, εκμεταλλεύονται αδυναμίες. Το κάνει αυτό η Κίνα για να πετύχει και να πάρει αυτό που θέλει. Ε, μιλάω για, χρησιμοποιώ τον όρο, ε, διπλωματία της, με βαθιές παγίδες, κρυφές παγίδες. Ε, η Σιλάνκα πριν από κάνα δύο μήνες παρέδωσε επίσημα το ε, λιμάνι του Χαμπαντότα για 98-99 χρόνια ε, για να πληρώσει το χρέος της. Στην πραγματικότητα είναι η παγίδα του χρέους. Οι Κινέζοι δανείζουν. Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι η, η Παγκόσμια Τράπεζα Κίνα, ούτε η Τράπεζα της Ασίας. Ε, μιλάμε για τιτλοποίηση ε, στρατηγικών ας πούμε, περιουσιακών στοιχείων κτλ. Για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Δεν θα μπω ας πούμε, σε ιστορικούς παλισμούς, τι σημαίνει ας πούμε, παράδοση νησιών για 99 χρόνια κτλ. δεν θέλω να κάνω παραλληλισμούς, ε, χρησιμοποιώ τα όσα είπε ο προηγούμενο ομιλητή. Ε, αν... ε, κάποια στιγμή ή μπορεί να διακοπεί αυτή η παρεμβατική στάση. Αλλά στη, αυτή τη φάση υπάρχει παρέμβαση. Υποτίθεται ότι δεν κάνει παρέμβαση, δεν δημιουργεί σφαίρε επιρροή και όχι οι γεμονικέ τάσει. Αυτό είναι το δόγμα τη, το επίσημο και καλά. Εδώ δεν υπάρχει συνέπεια με αυτό. Αυτή η αμφισημία είναι ένα άλλο στοιχείο κλασικό στην, ε, στο κοινωνιστικό αφήγημα και συμπεριφορά. Γίνεται επίτηδε. Είναι βολικό, είναι πρακτικό. Δημιουργείται μια, ένα νεφέλωμα πίσω από το οποίο ο καθένα φαντάζεται ότι θέλει. και απλώς συμπερδεύει, γιατί το αφήγημα είναι τελείως διαφορετικό από την πραγματικότητα. Αυτό βλέπουμε στη θάση της Νότιας Κίνας, στον Ειδικό Ωκεανό και συχνά οι αναλυτές χρησιμοποιούν ε, ιστορικά παράλ... ιστορικούς παραλληλισμούς για να δουν αν η προσέγγιση είναι μαχανιακή, αν είναι προσέγγιση τύπου Σουν αλλά είναι επιλεκτική και είναι πολύ δύσκολο να την καταλάβει κανείς. Επίσης είναι μια εξελισσόμενη ισχύς και αυτό είναι καλό και κακό. Είναι κακό γιατί σε ορισμένε περιπτώσεις ισχυρίζονται ότι κάποια μη στρατιωτικά λιμάνια δεν θα χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς. Ε, αλλά τελικά αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν, αλλάζει η πραγματικότητα γιατί δεν υπήρχε από την αρχή διαφάνεια. Και τελικά φτάνουμε σε μία... Σε, σε, σε δεδομένα που δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, σε πεπραγμένα. Τέλος πάντων, πάντως μαθαίνουμε και μπορεί η, δύναμη, η ναυτική δύναμη της Κίνας μπορεί να φτάσει σε ένα επίπεδο ρημότητας όπου θα είναι πολύ πιο εύκολο να την καταλάβει κανείς. Αυτή η εξελικτική θεωρία είναι ότι τελικά όταν μάθει κανεί αρκετά, οι Κινέζοι αν προκειμένου να μάθουν αρκετά, θα αρχίσουν να συμπεριφέρονται πιο υπεύθυνα. Ο θαλάσσιος ε, δρόμος του μεταξιού, όταν ξεκίνησε την, ε, το εγχείρημα αυτό η Κίνα ή την επέκταση αυτή, χρησιμοποίησε ε, το παραδείγμα του στρατηγού Σεν Κιέ του 15ου αιώνα για να τονίσει την ειρηνική, τον ειρηνικό σκοπό ας πούμε, της επέκτασης αυτής. Ε, μιλάμε για την τέχνη της συνεργασίας, αυτό χρησιμοποιούν. Υποτίθεται μια συνεργασία που είναι υποφελής για όλους. Διαφάνεια, γενεοδορία, ε, ασφαλές ε, εξωτερικό περιβάλλον. Ήδη το 15ο αιώνα κυνηγούσαν τους πειρατές. Υπάρχουν στοιχεία και αυτής της τάσης αλλά υπάρχουν και στοιχεία ε, της ε, στρατηγικής Σουν Τσου. Ε, το να χρησιμοποιήσεις αδυναμίες ε, και να κερδίσεις τον κόσμο χωρίς να δώσεις μάχη είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχεί τους υπόλοιπους. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν. Αλλάζει η στρατηγική ισορροπία στην, ε, στον Ειδικό Ωκεανό, στον Ειρηνικό. Βλέπουμε την, τα στοιχεία μιας τετραμερούς συμμαχίας Πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά. Βλέπουμε αυτή την οικονομική επιρροή που χρησιμοποιείται για να εξαγοραστεί η πολιτική θέληση πολλών χωρών και στην άμεση γειτονία της και στην άμεση γειτονία μας επίσης, Δυτικά Βαλκάνια, που είναι ένα από τα πρώτα μας μελήματα, αλλά και στην εσωτερική στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπάρχουν τέτοια θέματα και τέτοια τάσεις και επιπτώσεις λόγω προβλημάτων με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν ε, κανόνες ε, για την παγκόσμια τάξη. υπάρχει κίνδυνος για αυτούς τους κανόνες. Και το θέμα με τον θαλάσσιο ή τον χερσαίο ε, δρόμο του μεταξιού είναι ότι δεν υπάρχει διακυβέρνηση αυτού. Ο θαλάσσιος ε, κινέζικος, ε, συγγνώμη, ο θαλάσσιος δρόμος του μεταξιού, όμως σήμερα ο σημερινός, αυτός που οικοδομεί η Κίνα, είναι κινέζο-κεντρικός. Παλιά δεν ήταν αυτό το πράγμα ο δρόμος του μεταξιού. Αν η Κίνα θέλει να γίνει παγκόσμιος ηγέτης, θα πρέπει να έχει και την ικανότητα την ηγετική. Και, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να το δουν αυτό η Ευρώπη και οι υπόλοιπε δυνάμει και ίσω να δείξουν μεγαλύτερη δραστηριότητα και ενεργητικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον ε, κύριο Άντρου Σκόπελ από τη Rand Corporation. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να συμμετέχω στη σημερινή συζήτηση. Οι παρατηρήσεις που θα κάνω είναι προσωπικές, δεν εκπροσωπούν τη Rand Corporation ούτε τους χορηγούς της. Ο σκοπός της σημερινής μας συνάντησης είναι να κάνουμε μια προβολή της ισχύω. Τι ακριβώς είναι η προβολή ισχύω. Ένας ορισμός του Ευρωπαϊκού Υπουργείου Άμυνας είναι ότι είναι η ικανότητα ταχαίως και αποτελεσματικά να αναπτύσσει κανείς και να συντηρεί δυνάμεις σε διάφορες τοποθεσίες από τις οποίες έχουν αποσταλεί και στις οποίες επιχειρούν. Είναι είναι περίπλοκος ο ορισμός, αλλά καταλαβαίνετε. Για ποιο λόγο λοιπόν πρέπει η Κίνα ή θέλει η Κίνα να κάνει μια προβολή της παγκόσμιας στρατιωτικής της ισχύω. Από το έγγραφο του 2015 που εξέδωσε ε, το Υπουργείο Άμυνας της Κίνας είναι, προκύπτει ότι είναι η εξασφάλιση των ε, εξωτερικών συμφερόντων, των υπερπόντιων συμφερόντων της Κίνας, ε, στο εξωτερικό δηλαδή. Ποια, ποια είναι αυτά τα συμφέροντα. Ενέργεια, πόροι, στρατηγική δρόμη μεταφοράς, ε, θεσμικά όργανα, προσωπικό και πολίτες της που βρισκόνται στο εξωτερικό. Τα συμφέροντα της Κίνας λοιπόν έχουν ολόνα και μεγαλύτερη σημασία και εμφανίζονται ολόνα και περισσότερο σε επίσημα κρατικά έγγραφα. Και αυτά όπως είπα περιλαμβάνουν και τους πολίτες της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας που ταξιδεύουν ή ζουν στο εξωτερικό και τις επιχειρήσεις της Κίνας, βεβαίως, που βρίσκονται στο εξωτερικό. Η ουσία όλων αυτών είναι βεβαίως οι άνθρωποι και τα πράγματα. Σε όλο τον κόσμο ζουν πλην της Κίνας, δηλαδή 5 εκατομμύρια πολίτες της ε, Κίνας, ένα εκατομμύριο είναι από αυτό στην, ε, στην Αφρική και μισό εκατομμύριο περίπου στη, στη Μέση Ανατολή. Επίσης, η Κίνα έχει κάνει επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλο τον κόσμο. Ο αριθμός των πολιτών της και το ύψος των ε, εξωτερικών επενδύσεων της Κίνας θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια στην πορεία και της ανάπτυξης αυτής της πρωτοβουλίας για, την, για δρόμο του μεταξιού που συζητούμε εδώ σήμερα και που ακούσαμε πολλά γι' αυτό. Αυτά τα φιλόδοξα σχέδια της Κίνας αλλά και γενικότερα οι σχεδιασμοί της χώρας ε, στον Ειρηνικό ωκεανό και στον Ινδικό ωκεανό έχει, έχουν προκαλέσει μια μεγάλη συζήτηση για το, εντός της χώρας για το πώς ακριβώς μπορούν να προστατευτούν και να εξασφαλιστούν τα συμφέροντά τους στο εξωτερικό. Μία από τις ε, βασικές επιλογές ε, της Κίνας ε, μάλλον όχι. Είναι πέντε οι επιλογέ που έχει η Κίνα. Έτσι όπω τι έχω κατηγοριοποιήσει εγώ θα σα τι παρουσιάσω. Λοιπόν, πρώτη επιλογή για την προστασία των προσωπικών ε, των, ε, συμφερόντων, των εθνικών συμφερόντων είναι στο να μην, στο να μην τηρείται κανένας κανόνας για παράδειγμα αξιοποιώντας τις ικανότητες άλλων χωρών. Η Κίνα, για παράδειγμα, εδώ και πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, βασίζεται στις ικανότητες των ΗΠΑ για την, ε, για την περιπολία και την εξασφάλιση, της, την προστασία της ασφάλειας σε μια σειρά από θαλάσσιες περιοχές, όπου η ίδια η Κίνα δεν έχει συμβάλει ποτέ. Η Κίνα βεβαίως ε, δεν θέλει να ε, βασίζεται ε, επαόριστον στον αλτρουισμό των ΗΠΑ. Δεύτερη επιλογή για την προστασία των υπερπρόντων συμφερόντων της είναι να επανεξετάσει τις συμμαχίες της και να ε, ενισχύσει τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις. Έπειτα από δεκαετίε όπου ακούγαμε ότι η Κίνα δεν συνάπτει συμμαχίε, τα τελευταία χρόνια το, το Πεκίνο συνεργάζεται όλο και πιο στενά στρατιωτικά με άλλε χώρε. Πλέον η Κίνα έχει μια ολόκληρη γκάμα σχέσεων με άλλες χώρες στον τομέα της ασφάλειας και ε, με πολύ απτά αποτελέσματα. Σε αυτές τις χώρες περιλαμβάνονται ε, το Πακιστάν για παράδειγμα, πολυμερείς σχέσεις και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην οργάνωση συνεργασίας της Σανγκάης, όπου βεβαίως συμμετέχει και η Ρωσία. Επίσης, κάποιες από τις σχέσεις της Κίνας με άλλες χώρες αρχίζουν να εμφανίζουν χαρακτηριστικά συμμαχίας. Τρίτη επιλογή για την προστασία των υπερπόντιων συμφερόντων της Κίνας και το ακούσαμε και σε μια προηγούμενη ε, παρουσίαση είναι η δημιουργία βάσεων στο εξωτερικό. Κάτι που μπορεί να είναι μπορεί να τις χτίσει μόνο σου ή να απλά να αξιοποιήσει λιμάνια άλλης χώρας. Αυτό είναι και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσο έχει προοδεύσει η σκέψη εντός της Κίνας σε σχέση με την προστασία των συμφερόντων της. Η Κίνα ε, πάντοτε ακολουθούσε μια πολιτική μη παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα άλλων χωρών. Και μάλιστα επέμενε για πολλές δεκαετίες η Κίνα ότι δεν έχει ε, αναπτύξει ε, στρατιωτικές δυνάμεις ποτέ σε άλλη χώρα. Ωστόσο, από το 2016 και έπειτα, με την ανάπτυξη ε, του ναυτικού της Κίνας ε, στον ε, στον κόλπο του Άντεν ε, έχει προκαλέσει μια μεγάλη συζήτηση για, το, για ενδεχόμενο αναπροσανατολισμό και ε, αλλαγή κατεύθυνσης. Υπάρχουν μια σειρά από λιμάνια και βάσεις ε, που φημολογείται ότι αποτελούν κινέζικες ναυτικές βάσεις στην πραγματικότητα όπως είναι το Γκουάνταρ στο Πακιστάν. Αν και εξ όσων γνωρίζω το Γκουάνταρ εξακολουθεί να είναι εμπορικό λιμάνι και όχι στρατιωτική ναυτική βάση. Τέταρτη επιλογή για την προστασία των υπερπόντιων συμφερόντων της Κίνας είναι η εξωτερική ανάθεση του τομέα της ασφάλειας. Να βασίζεται δηλαδή η Κίνα στην, ε, στην ε, ε, φιλοξενούσα χώρα ή και σε ιδιωτικές εταιρείες προκειμένου να εξασφαλίζουν και να προστατεύουν τα συμφέροντα των Κινέζων στο εξωτερικό. Έπειτα από το συμβάν στο Ισλαμαμπάν το 2017 η χώρα αυτή, το Πακιστάν, ε, αναγκάστηκε να δημιουργήσει ειδική δύναμη αστυνομική για την προστασία των πολιτών της Κίνας στο έδαφος του Πακιστάν. Σε άλλες χώρες ε, η Κίνα έχει αναθέσει ε, ιδιωτικά συμβόλαια σε εταιρείες προκειμένου να προστατεύονται τα, τα κινέζικα συμφέροντα. Πέμπτη επιλογή για την προστασία των συμφερόντων της Κίνα είναι βεβαίως η ενίσχυση και η διεύρυνση των ικανοτήτων προβολής παγκόσμιας ε, ισχύω της Κίνα ε, σε άλλες χώρες. Συγκεκριμένα αναφέρομαι ε, στην, στην αεροπορία και στο ναυτικό. Ο εξυγχρονισμός του στρατού στην Κίνα έχει ήδη θέσει ε, το ναυτικό της, της, της χώρας αυτής σε νέες βάσεις, αλλά αναμένονται και επιπλέον εξελίξεις, ε, όχι μόνο στο ναυτικό, αλλά και στην ακτοφυλακή της χώρας. Το ναυτικό λοιπόν του Λαϊκού Στρατού της Κίνας αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να προβάλλει ε, ιδιαίτερη ισχύ πέραν της Ανατολικής Ασίας. Ε, υπάρχουν ορισμένες ναυτικές βάσεις και ορισμένα σημεία σημαντικά στον Ειρηνικό και στον ε, Ινδικό ωκεανό, αλλά ε, εξακολουθεί το ναυτικό της να είναι ανεπαρκές προκειμένου από μόνο του τουλάχιστον να προστατεύσει το σύνολο των παγκοσμίων συμφερόντων της Κίνας. Το αεροπορικό πρόγραμμα της Κίνας δείχνει την ξεκάθαρη επιδίωξη της Κίνας ε, για επίδειξη ε, δύναμης και σε αυτόν τον τομέα. Όμως μέχρι στιγμής η Κίνα έχει μόνο ένα έχει μόνο ένα ε, λειτουργικό αεροπλανοφόρο. Αυτή τη στιγμή ναυπηγείται και το δεύτερο, αλλά δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία, σε υπηρεσία θα χρειαστούν κατά πάσα πιθανότητα χρόνια έως ότι το Πεκίνο καταφέρει να διεκπεραιώνει, ε, να εκτελεί ναυτικές στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως αυτές που έχουμε συνηθίσει από τις ΗΠΑ. Οι ε, ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν χερσαίες δυνάμεις αλλά και ναυτικό και την αεροπορία θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια έως ότου καταφέρει η Κίνα να εκτελέσει. Κάποιοι εκτιμούν ότι ε, η Κίνα θα προβεί σε μαζικές ε, προσλήψεις στο ναυτικό της. Κάτι που θα της επιτρέψει ε, να κάνει ναυτικές επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά αυτά είναι οι κασίες επί του παρόντος τουλάχιστον. Οι αλλαγέ πάντω και οι μεταρρυθμίσει στο ναυτικό τη Κίνα σε κάθε περίπτωση αξίζει να τι ε, παρακολουθήσουμε. Οι δυνάμει ε, του Κινέζικου στρατού επίση ε, αρχίζουν και προβαίνουν σε προβολή ισχύω και στην περιφέρεια τη χώρα. Όλο ένα και περισσότερα. Όλο ένα και περισσότερα στρατεύματα είναι στη διάθεση ανα πάσα στιγμή του Υπουργείου Άμυνας της Κίνας προκειμένου να τεθούν ή να αποσταλούν σε συγκεκριμένες στρατηγικές επιχειρήσεις. Και αυτό ένα και πιο μακριά από την υπηρετική Κίνα, ε, κάτι όμως που βεβαίως αυξάνει και το κόστος ε, για τον Κινέζικο στρατό. Μια ε, εναλλακτική θα μπορούσε να είναι να προβεί στην τελειοποίηση της, του εναέριου ανεφοδιασμού καυσίμου για την, ε, για την Κίνα. Η ικανότητα του κοινωνικού στρατού λοιπόν ε, στο να χρησιμοποιεί διάφορες τέτοιες πλατφόρμες ε, περιορίζεται από τις, τους περιορισμένους πόρους που έχει εκτός κινέζικων συνόρων. Ακούσαμε για το Τζιμπουτί όπου υπάρχει ένας κόμβος επιμελητίας που προς το παρόν αποτελεί ένα ελαφρύ ίχνος, ελαφρύ σε σχέση με το ίχνος ε, του Αμερικανικού στρατού στον κόσμο, ε, το οποίο είναι πολύ πιο ε, έντονο. Όταν λέμε ελαφρύ ίχνος, μιλάμε ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις για εκατοντάδες Κινέζους που δουλεύουν σε όλη την αλυσίδα επιμελητίας. Η Κίνα, λοιπόν, έχει υιοθετήσει ένα μείγμα αυτών των ε, παραπάνω επιλογών που σας παρουσίασα. Ε, κάνει λίγο απ' όλα. Συμμαχίες, στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις, αναθέτει εξωτερικά, ε, παραβιάζει και κανόνες ή χρησιμοποιεί τους πόρους ε, άλλων χωρών για να εξυπηρετεί στα δικά της συμφέροντα. Συνοπτικά λοιπόν η Κίνα θα εξακολουθήσει να είναι υπολογίσιμη, ισχυρή περιφερειακή δύναμη που θα μπορεί να προβάλλει την στρατιωτική της ισχύ, ιδίως στη γειτονιά της, στον Ειρηνικό και στον Ινδικό ωκεανό. Και οι ικανότητες της αυτές ε, μάλλον θα βελτιωθούν τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, πέραν αυτής της ε, περιφέρειας του ε, Ειρηνικού και του Ινδικού, κατά πάσα πιθανότητα η Κίνα δεν θα μπορέσει να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, τουλάχιστον έως τα μέσα της δεκαετίας του 2020. Με τη δύναμη κρούσης ε, κατά της ε, πειρατείας αλλά και με την δυνατότητα της Κίνας που επέδειξε στη Λιβύη για την εκένωση των πολιτών της ε, το 2011 ε, οι προβολές του κινέζικου στρατού μέχρι στιγμής εμφανίστηκαν μόνο μία φορά η κάθε μία. Και αυτοί ε, στη Λιβύη ε, χρησιμοποιήθηκαν 76 αεροσκάφη για την εκένωση Κινέζων πολιτών κατά την κρίση της Λιβύης. Τέσσερα από αυτά τα, ε, αεροσκάφη ήρθαν από την Κίνα. Κάποια ήρθαν από άλλες χώρες, από αεροπορικές βάσεις της, της Κίνας στην Αφρική και όλα αυτά για έναν σχετικά μικρό αριθμό Κινέζων πολιτών. Ήταν εντυπωσιακό, ήταν μια επίδειξη δύναμη, αλλά μην θεωρήσετε ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί η Κίνα να το κάνει καθημερινά. Σε κάποιες ή και στις περισσότερες περιοχές ε, του κόσμου ε, η Κίνα παρά την ενισχυμένη της οικονομική δύναμη ε, θα εξακολουθήσει διπλωματικά να έχει πολύ μικρότερη σημασία από την οικονομική σημασία δηλαδή και στρατιωτικά ακόμα μικρότερη. Βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε ε, μια πιο ορατή παρουσία των κινέζικων στρατευμάτων σε διάφορες περιοχές του κόσμου, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, ε, στην πορεία της ε, επόμενης δεκαετίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε αξιότιμη κύριε. Πριν να δώσω το λόγο στα μέλη εδώ για την γενικότερη συζήτηση, να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, τον κύριο Φράνκαρ. Έγγελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν με είχα μετρήσει πρόσφατα αεροπλανοφόρα της Κίνας, δεν ξέρω ακριβώς ο αλλά μια χώρα που χάνει ε, μισό εκατομμύριο ανθρώπους στον πόλεμο της Κορέας. Και αυτή ήταν εκτίμηση των ΗΠΑ όταν είχαν το 1 τρίτο των κατοίκων που έχουν σήμερα. Μπορεί να βρει τους, ε, τα πλοία που έχει σήμερα, πάρει τα πλοία που έχει σήμερα και του ανθρώπους που έχει σήμερα και να πάει να πάρει, καταλάβει την Ταϊβάν. Κάποια πράγματα έχουν αλλάξει την τελευταία δεκαετία ούτως ή άλλως. Το γνωρίζουμε στις επαφέ μας μαζί τους. Δεν έχουν τα πράγματα όπως είχαν και πιθανώ θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Ορισμένοι από εμά ε, έχουμε προσκληθεί προσκληθήκαμε τι τελευταίε μέρε του Δεκεμβρίου στο Παγκόσμιο Φόρουμ ε, στο Καθολικό Φόρουμ των Πολιτικών Κομμάτων, μια περίεργη πρωτοβουλία όπου συναντήσαμε ε, με τριοπαθείς δημοκράτες ε, όπως τον Σαν μέχρι και εκπροσώπους του, των Ρεπουμπλικανών των ΗΠΑ. Και όταν όλα είχαν τελειώσει, μας έδωσαν ένα χαρτί, 7-8 σελίδες, ένα έγγραφο, που υποτίθεται έπρεπε να επικυρώσουμε το ονόμαζαν πρωτοβουλία του Πεκίνου που συνίστατο σε ένα πολύ παράξενο ύμνο για το 19ο Κογκρέσο του Κόμματος και τον εξαιρετικό πρόεδρο, το συνέδριο του Κόμματος και τον ε, πρόεδρο, τον εξαίρετο πρόεδρο Σι Τζιμπινγκ. Σας διαβεβαιώ ε, ότι κανένας που εκπροσωπούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ε, έβαλε την υπογραφή του στο έγγραφο αυτό, αλλά τώρα φαίνεται ε, ότι οποιοδήποτε πάει στην Κίνα πρέπει να τους εγκρίνει με αυτόν τον τρόπο. Ε, ότι πάμε εκεί δηλαδή και πρέπει να τους ε, καταβάλουμε τα σέφη και αυτό δεν πρέπει να μας πλανά. Βλέπουμε, φαίνεται ότι σχεδιάζουν τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουν πάει μόνο στο Τζιμπουτί. Στο Τζιμπουτί, αλλά στην Αφρική και μόνο υπάρχει και ε, ένα λιμένας ε, μεγάλο στο άτομο και πρίncιπε πολλών εκατομμυρίων επένδυση που δεν ήθελε να δώσει η Ταϊβάν. Ταϊβάν δεν ήθελε να χτίσει βάση εκεί, αλλά εκείνα ναι. Καθοδόν ε, για την άλλη βάση που βρίσκεται στι Αζόρε, που δημιουργεί πολλά προβλήματα τώρα σε συνομιλητέ από την Πορτογαλία. Και πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο είναι ευχάριστο για μας και κατά πόσο μας κάνει να νιώθουμε άνετα το να περιβαλλόμαστε από κινέζικες βάσεις που δεν έχουν καμία λογική να υπάρχουν εκεί, δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τη μία ζώνη, μία οδό, μία ζώνη, ένα δρόμο, η Κίνα. Η Κόσκο βέβαια έτσι, αλλά πρόκειται για την Κίνα ουσιαστικά. Όπως και η τράπεζα έξω στην Αφρική είναι Κίνα. Η Κόσκο δεν αγόρασε τα λιμάνια της Αθήνας και για το τίποτα ήταν οι πρώτες φυσικές βάσεις πρώτα για τα προϊόντα της κόσμο και μετά για όλα τα άλλα. Τη μορφή 16 16-1 δεν την επινοήσε η Κίνα για, χωρίς λόγο και παρότι θεωρώ ότι είναι ντροπή ότι 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν με αυτή την απάτη απλά διότι τους υποσχέθηκαν κάποια προϊόντα 3 ε, εκατομμύρια ευρώ κάποια πράγματα Τρία ε, και φαίνεται ότι λειτουργεί το πράγμα διότι στις τελευταίες ψηφοφορίες των ΗΠΑ ε, η ε, επίσημη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπήρχε πλέον και η Ελλάδα και η Ουγγαρία για περίεργους λόγους δεν ψήφιζαν μαζί με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορούσε την Κίνα και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα συνεχιστεί και ότι τελικά όλο και περισσότερες χώρες θα ψηφίζουν αντίθετα από το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επιτρέπει και παρέχει και ε, υποστήριξη υποδομών στο 16.1 σε αυτό το δίκτυο. Αν θέλουμε εμείς να έχουμε μια ενιαία πολιτική για την Κίνα καθημερινά και αυτοί θα πρέπει να έχουν μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Αν μας έπαιρναν σοβαρά φυσικά, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Αν εμείς παίρναμε τον σοβαρά, θα πηγαίναμε να δούμε τι συμβαίνει ε, στο 19ο συνέδριο και από τότε που υπήρχε ο Σιντζιμπίνγκ βλέπουμε ισχυρή συγκέντρωση εξουσιών στα χέρια ενό ανθρώπου στην Κίνα που υπάρχει από τι αυτοκρατορικέ ημέρε. Ε, Ισχυρότερο από το ΜΑΟ πιθανότητα, διότι σίγουρα υπάρχει καλύτερη οργάνωση. Ο ΜΑΟ είχε τι χαοτικέ του στιγμέ και τι ε, ε, τυχαίε. Ε, δεν νομίζω ότι είναι τίποτα τυχαίο αυτή τη στιγμή στην Κίνα. Και επίσης είμαι πεπισμένος ότι η Κίνα δεν θα συνεχίσει να υλοποιεί τον δεκαετή κανόνα για τη μεταβίβαση εξουσία όταν θα τελειώσει η θητεία του Προέδρου Σι. Φανταστείτε τώρα, σκεφτείτε πόσο χρονών είναι. Είναι στα, στα 60, 60 τόσων. Δηλαδή μπορεί να παραμείνει για άλλα 15 χρόνια. Μέχρι τότε αυτός και όλη η λογική που οικοδομείται αυτή τη στιγμή γύρω από τον Πρόεδρο της Κίνας θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει την ιστορική αποστολή και φιλοδοξία του κινέζικου λαού, δηλαδή πρώτα απ' όλα να αποκαταστήσει την ιστορική ενότητα της ε, ε, χώρα του, τη Πατρίδα. Του. Δεν του ενδιαφέρει ότι για χιλιάδε χρόνια ε, κανένας Κινέζος δεν είχε βάλει το πόδι του στην Ταϊβάν. Αυτό που του ενδιαφέρει είναι ότι αυτή τη στιγμή του ενδιαφέρει ότι η Ταϊβάν πρέπει να ξαναγίνει κομμάτι τη Κίνα. και θα γίνει και μπορεί να ρηψοκινδυνεύσουν άλλο ένα τέτοιο ε, σχήμα. Όπως ήταν, λίγο ουσιαστικά συμπεριφορά Τραμπ. Ε, αλλά κατά τα άλλα έχουν εξαγοράσει τόσο κόσμο σε όλο τον κόσμο που κανείς δεν πρόκειται να παραπονεθεί. Και απλά θα κοιτάμε αλλού και θα πούμε ε, ούτως ή άλλως δεν είχαμε αναγνωρίσει την Ταϊβάν. Έτσι δεν είναι. Είμαι πεπισμένος ότι η Κίνα δεν πρόκειται να εισβάλλει στο Περού, στον Καναδά ή στην Ιρλανδία αύριο. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι Πρώτα το Χονγκ Κόνγκ, μετά η Ταϊβάν. Θα δούμε για τη Μογγολία, θα το συζητήσουμε αργότερα. Πόσο καιρό θα διατηρήσουμε την ειρήνη στην νότια Συνική θάλασσα, όσο εμείς τους επιτρέπουμε να ε, υλοποιούν ε, προσβλητική πολιτική, ε, να βάζουν σταθμούς παντού, που σε μέρη που δεν ήταν ποτέ κινέζικα και που εμείς δεχόμαστε, πέραν της διεθνούς διαιτησίας. Καθόμαστε και κοιτάμε αλλού όταν αυτά συμβαίνουν. Αυτό λοιπόν συνεχίζεται όσο όλοι διστάζουμε, όποιος τολμήσει να τους προκαλέσει θα τον προκαλέσει και εκείνα. Και ε, όπως φαίνεται θα συνεχίσουν αυτή τη μέθοδο διότι όπως ε, υπόθηκε και εδώ μπορεί να μην μπορούν να, να κάνουν μια τεράστια παγκόσμια εισβολή αλλά μια μικρή κίνηση στις δικές τους θάλασσες γύρω από την Κίνα δεν τους είναι και τόσο δύσκολο. Αυτό λοιπόν είναι άλλο ένα πρόβλημα το Χονγκ Κόνγκ επηρεάστηκε πρώτο και η Ταϊβανή μπορεί να είναι η επόμενη. Πριν από 10 χρόνια το Hong Kong. οικονομικά ήταν τόσο σημαντικό μέσα στην Κίνα Δεν υπήρχε άλλη πόλη 6-7 εκατομμυρίων που να μπορούσε να συναγωνιστεί το Hong. Κόνγκ. Οπότε το άφηνα στην ησυχία του. Αλλά τώρα το έχουν ξεπεράσει τόσε πολλέ άλλε πόλει στην Κίνα, το Σεντζέν πρώτα απ' όλα, στην άλλη πλευρά των συνόρων ουσιαστικά, που δεν χρειάζεται το Hong Kong τόσο πολύ. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα αντέξει. Και η Ταϊβάν πριν από 10-20 χρόνια θα μπορούσαν να την είχαν ε, ε, κατακτήσει. Αν την καταστρέφαν θα μπορούσαν να γίνει δική τους. Αλλά τότε ήταν ανταγωνιστή της Κίνα σήμερα. δεδομένη της οικονομικής ε, δύναμης της Κίνας η Ταϊβάν είναι αναλώσιμη και αυτό είναι κακό νέο για τους Ταϊβανού που είναι μόλι 23 εκατομμύρια. Είναι ένα μεσαίο κράτο μόνο τη Ευρωπαϊκής Ένωση μικρό κράτος ε, και αυτό μας ειδοποιεί για πράγματα που μπορεί να συμβούν. Είμαι πεπισμένος ότι η Κίνα είναι αποφασισμένη να κάνει παραπάνω από ό,τι εμείς υποθέτουμε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να φαίνεται ήρεμη, καθησυχαστική, κατά καιρούς αλλά και αυτό αλλάζει. Τα γεγονότα έχουν αλλάξει εδώ και καιρό. Thank you, sir. Yes, Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έχουμε μια μεγάλη ομάδα ευρωβουλευτών ε, που υποστηρίζουν την Ταϊβάν. Έχουμε ε, συζητήσει το θέμα αυτό και θα το συζητήσουμε και αργότερα σήμερα. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπράφκα Σουίτσα που είναι αντιπρόεδρος της ΑΦΕΤ, της Επιστροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Άκουσα αυτά που είπε ο κύριος Έγγελ. Γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω για την παγκόσμια διάσταση σε σχέση με αυτά που είπε η, η αναλύτρια η Εύα παίσοβα θέλω να σχολιάσω τα εξή. Εσείς αναλύσατε την θαλάσσια ισχύ της Κίνας. Μια συγκεκριμένη ερώτηση έχω να κάνω για την Ταϊβάν. Αναφερθήκατε και στην αεροπορία. Δεν ξέρω αν ξέρετε διάφορα πρόσφατα στοιχεία. Ξέρετε τα εξή θα σας πω. Η πολιτική αεροπορία της Κίνας μονομερώς ανακοίνωσε στις 4 Ιανουαρίου του 2018 ότι θα ε, ενεργοποιήσουν χωρίς πρώτερη ε, διαβούλευση με την Ταϊβάν ε, τον κανόνα 503, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, για τέσσερις δρόμους, πολύ κοντά στην στους ενέριους δρόμους της ε, Ταϊβάν μπορεί να παρέμβει με την πολιτική αεροπορία της Ταϊπέη ε, και το ΦΥΡ ε, Ταϊπέη. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν θεωρεί ότι αυτό είναι μολομερής κίνηση από την Κίνα, μία μη υπεύθυνη κίνηση που επηρεάζει την πολιτική αεροπορία της Ταϊβάν και τα στενά Ταϊβάν-Κίνας παρεμβαίνει στους δρόμους που χρησιμοποιεί, στους ε, εναέριους δρόμους που χρησιμοποιεί, η πολιτική αεροπορία κτλ. Και αυτό ουσιαστικά ε, απειλεί στην Ανατολική Ασία την ειρήνη και σταθερότητα και δεν συνάδει με τις απόψεις που εκφράζουν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις εκθέσεις του για την εφαρμογή της ΚΠΑ και τις απόψεις που εκφράσαμε πέρυσι για το Χονγκ Κόνγκ. Ήμουν σκιώδης εισηγήτρια. Την έκθεση αυτή την υιοθετήσαμε το Δεκέμβριο του 2017. Ποια είναι η άποψή σας. Έχουμε θέση γι' αυτό. Τι έχετε να πείτε για αυτό το θέμα. Thank you. Uh, Claire Moody, Vice uh, Chair of SEDA. Αντιπρόεδρος της uh, SEDA, Claire uh, Moody. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήρθα νωρίτερα. Θέλω να ακούσω την απάντηση που θα δώσετε στα όσα ακούσατε μόλις τώρα από την προβαλή σας. Το δικό μου συγκεκριμένο ερώτημα ε, αφορά τα σχόλια του κύριου Σκόμπελ. Μιλάμε για την προστασία του προσωπικού, των ανθρώπων δηλαδή και του προσωπικού. Δεν ξέρω αν το κάλυψαν οι προηγούμενοι ομιλητέ πριν φτάσω εγώ. Ζητώ συγγνώμη αν έγινε αυτό αν έγινε κάτι τέτοιο, αλλά θεωρούμε ότι η Κίνα έχει μία αμυντική στρατιωτική α, στρατηγική ή πέρασε σε επιθετική φάση. Και κάτι συναφές. Σε άλλες συγκρούσεις που ξέρουμε, βλέπουμε ότι γίνονται πόλεμοι για αντιπροσώπου. Ε, μπαίνουν και επισέρχονται και συμμετέχουν ας πούμε σε συγκρούσεις άλλων κρατών κάποιες χώρες. Γίνονται πόλεμοι δια αντιπροσώπου. Στην κοινωνική πολιτική βλέπετε για στοιχεία πολέμου, πολέμου δια αντιπροσώπου. Και κάτι άλλο. Μπορεί να καλύφθει και το συγγνώμη αν ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο μέλημα. Ε, η κυβερνοδραστηριότητα της Κίνας. Μεγάλο μέλημα, μεγάλο πρόβλημα. Τι γίνεται με τους κρατικούς φορείς που κάνουν ε, κυβερνοπαρεμβάσεις σε όλους τους τομείς. Κοιτάξτε, τις παρεμβάσεις σε υποδομές, αλλά και σε άλλους τομείς. Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο κ. Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Αυτές που μας δείξατε μάλιστα εδώ στην οθόνη, δεν ξέρω αν θα μπορούσατε ενδεχομένως να μας τις στείλετε ήταν πολύ ενδιαφέρον κάτι τέτοιο. Η μία παρουσίαση λοιπόν έδειξε κάποια στιγμή έναν μεγάλο χάρτη με διάφορες θέσεις όπου έχουν ήδη παρουσία οι Κινέζοι. Εγώ όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με την εξωτερική πολιτική ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 80. Εκεί ε, τότε ο τίτλος ήταν «Το δίχτυ της κόκκινης αράχνης» και έδειχνε σε μια πορεία χρόνου πόσο μεγάλωνε η επιρροή στην Αφρική, στην, στην Ασία της Σοβιετικής Ένωσης. Και η πρόβλεψη τότε ήταν, ε, ό,τι και αν ήταν, πάντως διαψεύστηκε. Γιατί δεν υπολόγιζαν εκείνες οι εκτιμήσεις έναν πολύ σημαντικό ε, παράγοντα, το ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν μια μονοκομματική δικτατορία ε, που είχε έναν και νέο στρατό και όταν κατέρευσε η χώρα κατέρευσε μαζί της και ο στρατός. Φυσικά η Κίνα έχει πολύ ισχυρή οικονομία αλλά δομικά εξακολουθεί να είναι μια μονοκομματική δικτατορία. Δεν ξέρω αν αυτό το στοιχείο έχει συνυπολογιστεί στις ε, εκτιμήσεις και τις προβλέψεις μας. Γιατί εγώ θέλω να πω ότι παρά την οικονομική του ισχύ εξακολουθούν να είναι ένα μονοκομματικό κράτος και από αυτή την άποψη δεν έχουν επαρκείς μηχανισμούς λήψη αποφάσεων, κατάλληλους μηχανισμούς ε, λήψη αποφάσεων, ε, ακόμη και εντό της χώρας, της επικράτειας δηλαδή της χώρας, υπάρχουν και εσωτερικές ε, ε, ε μεταβλητές, άγνωστοι ε, που δεν, μας, δεν πρέπει να μας οδηγούν απαραίτητα στο συμπέρασμα ότι θα μπορούν για αενάως να διατηρούν αυτή την ναυπηγική του ισχύ, την, ε, τον έλεγχο ακόμη και των ίδιων τους των ε, περιφερειών. Υπάρχει αυτό το δομικό, εγγενές, διαρθρωτικό έλλειμμα στην, ε, στην Κίνα λοιπόν και δεν ξέρω αν έχει συνυπολογιστεί επαρκώς όταν σκιαγραφούμε τη συνολική εικόνα για αυτή τη χώρα. Και καθώς μας απασχολούν και τα ζητήματα έρευνας και στρατιωτικών εικονότητων, πέραν από τους αριθμούς του προϋπολογισμού της Κίνας για τις στρατιωτικές δαπάνες, έχουμε ε, συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά τις έρευνες που εκπονούν οι Κινέζοι στον αμυντικό τομέα. Υπάρχουν στατιστικά δεδομένα τα οποία έχουν έρθει στην ε, ε, υποπέσει στην αντίληψή μας, τα έχουμε συλλέξει αυτά για να μπορέσουμε να, να σχηματίσουμε και μια συνολικότερη εικόνα για το μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Φρανσβουλίκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ομιλητές. Θα ήθελα να εκφράσω ε, την άποψή μου για κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι στο μέλλον καλό είναι να υπάρχει πάντοτε και ένας εκπρόσωπος της χώρας την οποία συζητούμε. Σήμερα, για παράδειγμα, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε και την κινέζικη θέση από το Κινέζικο Ίδρυμα Διεθνών Σχέσεων, Διεθνών Μελετών, ε, Άμυνας, Ασφάλειας μαζί και βεβαίως ε, την άποψη των Αμερικανών. Κάτι τέτοιο θα μας οδηγούσε σε μια καλύτερη εικόνα, πιο ισορροπημένη. Ε, είναι λοιπόν δεδομένο ότι η Κίνα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην άμυνα και στην ασφάλεια, αλλά και ω προ την ε, εθνική της οικονομία. Και το ερώτημά μου είναι ε, ιδίως προς, τους, ε, προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση είναι για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με την Κίνα βάσει των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων. Γιατί υπάρχει τέτοια στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Ο κύριος ε, Σκόμπελ δεν είναι εκπρόσωπος του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών και ούτως ή άλλως ε, η ΕΠΑ είναι σύμμαχος ε, των περισσότερων ε, ευρωπαϊκών χωρών γιατί ανήκουν στο ΝΑΤΟ οπότε δεν είναι αυτό προτεραιότητα κυρία Ανδρικέα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους ομιλητές μας για τη συμβολή τους πρέπει να πω ότι αυτή τη βδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται να επισκιάζονται τα πάντα από την Κίνα και, τη σχετική της, ε, και την παγκοσμία της στρατηγική γιατί κοιτάξαμε το μηχανισμό ελεγχού των ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε ήδη συνέπειες, παρατηρούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη μας διάφορα αποτελέσματα. Εγώ είμαι από τη Λιθουανία. Ξέρετε, βρισκόμαστε πάνω στην Βαλτική και πολλοί συμπατριώτες μου θεωρούν ότι η Κίνα Έχει λόγο να αγοράσει η Κίνα εκεί ένα λιμάνι σε μια τόσο μικρή χώρα. Δεν βλέπουν καν που είναι οι Κινέζοι. Είναι στην άκρη όμως το λιμάνι, ε, εκεί ενός ε, από τους διαδρόμους ε, τους εμπορικούς και ο Πρωθυπουργό μας πρόσφατα κλήθηκε να έρθει στη Βουδαπέστη για να συναντήσει τον Κινέζο Πρωθυπουργό και η Λιθουανία τελικά υπέγραψε το πρωτόκολλο διατύπωση προθέσεων που αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής ομπόρ. Είμαστε λοιπόν κομμάτι αυτού του μεγάλου παιχνιδιού. Είμαστε πιόνι αυτού του παιχνιδιού και μας ανησυχούν οι συνέπειες. Ήθελα να αναφέρω και την κατάσταση στην Αποανατολή, η οποία έχει αλλάξει δραματικά τελευταία. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν τη Κορέα και φυσικά και το ε, ε, ενίσχυση του στρατιωτικού προφίλ της Κίνας όπως αναφέρατε ε, σήμερα στην περιφέρεια, στην περιοχή αυτή καθώς και η πρόσφατη μονομερής της απόφαση να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί ε, αμφιλεγόμενες αμφιλεγόμενους αεροδιαδρόμους έξω από την Ταϊβάν. Αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας του 2015. Δείχνει ότι η Κίνα έχει πρόθεση να εντείνει την ε, εξουσία της με μη στρατιωτικά μέσα στην περιοχή. Αυτό φυσικά δημιουργεί σοβαρές ε, ανησυχίες. Επειδή φαίνεται να συγκαλύπτει έτσι η Κίνα τις προθέσεις της προς την Ταϊβάν υπό το πρόσχημα της ε, πολιτικής αεροπορίας. Εάν η Ταϊβάν προσπαθήσει να αποκτήσει ανεξαρτησία και ξέρουμε ότι ο Ταϊβανός πρόεδρος το κόμμα το οποίο έχει υποστηρίξει την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Ξέρουμε τι υπόθηκε στην προεκλογική εκστρατεία. Ε, η κινέζικη κυβέρνηση ωστόσο έχει υποσχεθεί να χρησιμοποιήσει ε, στρατιωτική δύναμη και έχει αυξήσει τις περιπολίες ε, στρατικών αεροσκαφών κοντά στην Ταϊβάν και των βομβαρδιστικών. Η Ταϊβάν εντείνει τις προσπάθειές της η Κίνα εντείνει τις προσπάθειές της για να απομονώσει την Ταϊβάν από τις πολυεθνικές ε, που ε, έχουν δραστηριότητες στην Ταϊβάν, την Delta Airlines, την Marriott, ε, τις ζητούν να αφαιρέσουν την Ταϊβάν από την από το κατάλογο χωρών στις ιστοσελίδες τους. Έχω μερικές ερωτήσεις λοιπόν προς τον κύριο Μάνη. Μα ναι, πρώτα απ' όλα, ποια είναι η αντίδραση τη ευρωπαϊκή Ένωση ε, στις αλλαγές αυτές. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερική δράση πώς αξιολογεί αυτέ τι εντάσει μεταξύ Ταϊβάν και Κίνα. Υπήρξε κάποια απόκριση, κάποια διπλωματικά μέτρα που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη γενικότερη παραβίαση της συμφωνίας, διότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι έχει νόημα ε, για την Ταϊβάν να, ανησυχεί για τι νέε διαδρομέ, τη διεθνού ε, και να ε, το αναφέρει στο ΙΝΙΑΤΑ, ε, στον Οργανισμό των Ηνωμένων που επιβλέπει τους διεθνούς ε, αεροδιαδρόμους αλλά ταυτόχρονα δεν είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών και δεν έχει επίσημους δεσμούς με την ΙΑΤΑ. Από το 2016 μάλιστα έχει απορριφθεί το καθεστώς παρατηρητή στην Ταϊβάν. Πώς βλέπετε τις δράσεις της Κίνας προς την Ταϊβάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θέλω και εγώ να κάνω κάποιες ερωτήσει. Ω τακτικό μέλος της ΕΝΤΕ αφορά θέματα που ανέφερε και την πρόφυγα Σουίτσο και η κυρία Αντροκένα σε σχέση με την πολιτική αεροπορία και, την πραγματική και, εικονική, και τον πραγματικό και εικονικό αποκλεισμό της Ταϊβάν ε, κάτι που υπονομεύει την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας σε σχέση με το, με το αεροδρόμιο της Ταϊπέη αλλά όχι και μόνο, αφορά και κάποιες ε, εσωτερικές πτήσεις στην Ταϊβάν οπότε η ερώτησή μου προς τον κύριο Μανέ ε, είναι η εξής ε, επειδή η απάντηση για όλες τις ευρωπαϊκές ε, αεροπορικές που πετάνε στην Ταϊπέη ε, ε, μετά από αυτή τη μονομερή δράση της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας υπονομεύεται έτσι η ασφάλεια ουσιαστικά Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό είναι βέβαιο και ξέρουμε ότι σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες αεροπορίας όταν έχουμε ε, Γειτονικέ ε, ζώνες πτήση θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία ε, να διασφαλίζονται ασφαλείς αεροδιαδρομοί για τις πολιτικές πτήσεις. Οπότε θεωρώ ότι εδώ πρέπει να παρέμβουμε και εμείς για να υπερασπίσουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. επικεντρωνόμαστε στην ε, ελευθερία της ε, των πλοήγησης των πτήσεων και επικεντρωθήκαμε και στην προβολή ε, της ισχύω και μιλήσαμε για, την, για το ναυτικό. Αναφέρθηκε και το ζήτημα της ασφάλειας και του πολέμου στον κυβερνοχώρο που έχει αναγνωριστεί πλέον από τον ΝΑΤΟ πρόσφατα ως ο επόμενος, το επόμενο πεδίο μάχης. Η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας ε, είναι στρατηγικός εταίρος μας, αλλά εμπλέκεται και αυτή με αυτό. Όχι μόνο η Ρωσική Ομοσπονδία. Και η ερώτησή μου είναι, μαθαίνουμε κάτι από την περίπτωση της Ταϊβάν όσον αφορά τα θέματα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο παρατηρείτε να υπάρχει κάποιο μοτίβο, κάτι επαναλαμβανόμενο, γιατί είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε. Κάτι ε, εξακολουθεί να είναι μια από τις μεγαλύτερες ε, δυνάμεις ε, στον τομέα της πληροφορικής παγκοσμίως και οικονομικά. Ίσως να υπάρχει κάτι που να μπορούμε να μάθουμε. Υπάρχουν και κάποια προβλήματα ε, λόγω του αποκλεισμού εκ μέρους της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Ε, δεν μπορεί η Ταϊβάν να ε, συμβάλλει ας πούμε στη δημοσιακή υγεία όταν υπάρχουν πανδημι... Ε, κίνδυνοι πανδημίες υπάρχουν απειλές δηλαδή προς την παγκόσμια υγεία και παγκόσμια ασφάλεια η χώρα έχει τεράστια εμπειρία σε θέματα δημοσίας υγείας Έχουμε και ως Πολωνοί συνδράμει σε αυτό. Υπήρξαν γνωστοί Πολωνοί επιστήμονες που συνέβαλαν σε όλο αυτό. Ίσως λοιπόν να μας αφορά το ζήτημα αυτό και ίσως να αξίζει τον κόπο να έχουμε και την Ταϊβάν να, να συμμετέχει στους οργανισμούς μας. Αυτό συμφέρει τους πολίτες της Ευρώπης, πιστεύω, ε, για θέματα παγκοσμίας ασφάλειας. Θα ήθελα να ακούσω τις σκέψεις για όλα αυτά. Όταν αναφερόμαστε στη Βόρεια Κορέα για την ασφάλεια της κορεατικής χερσονήσου και αυτό είναι κάτι ανησυχητικό για όλους μας. Υπάρχει τρόπος ε, να ασκήσουμε πίεση στη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Κύριε Φρουντζουλίτσα, ε, αυτός ε, ο στρατηγικός μας εταίρος ε, ε, πώς θα ασκήσουμε περισσότερη πίεση στην Βόρειο Κορέα για να υπονομεύσουμε τον πυρηνικό κίνδυνο από αυτό το καθεστώς του κίνημα. Αυτές ε, είναι τα ερωτήσει μου. Ας ε, αρχίσουμε με την ίδια σειρά. Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Μανέ, με τα κυρία Πέσοβα και με τον κύριο Σκόβολ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, Θα απαντήσω στην εξή ερώτηση. Κάποιος ευρωβουλευτής είπε ότι υπάρχουν και επιπλέον ίσως παράμετροι που δεν λαμβάνουμε υπόψη όταν αξιολογούμε την κινέζικη ισχύ της Κίνας και την προβολή της κινέζικης ισχύς. Αναγνώσα και στην ομιλία μου ότι η Κίνα έχει ικανότητες όλο και μεγαλύτερες, αλλά είναι σημαντικά να, σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας και να παράγοντα που είναι η γεωγραφία. Η Κίνα έχει αυτά που έχει. Αν λάβουμε υπόψη μας και τη, και τη γεωγραφία, μπορούμε να πούμε την γεωγραφική θέση της Κίνας ως ε, ιδιαίτερος αδύναμη. Είναι μια υπηρετική δύναμη κατεξοχήν ή κυρίως. Μπορεί να περιοριστεί και να εξουδετερωθεί εύκολα και συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κίνα στην προβολή της αυτή είναι εδώ βρίσκεται... Από, μπορεί να εξουδετερωθεί από τους συμμάχους, ε, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, Αυστραλία, Σιγκαπούρη και την Ινδία που είναι με, πέρα από τα 200 μίλια των χωρικών υδάτων της. Το είπε και ο κύριος Σκόμπελ αυτό. Οι επιχειρήσεις ε, οι μακρινές είναι εξαιρετικά δύσκολες για τη χώρα αυτή και θα παραμείνουν δύσκολες για τις επόμενες τρεις, τέσσερις ή πέντε δεκαετίες. Και ένας τεράστιος στρατιωτικός προπολογισμό δεν αλλάζει τα γεωγραφικά δεδομένα. Με ρωτήσατε η, ποια είναι η συνεργασία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας είναι το, μια συνεργασία που τώρα γεννάται, κυρίως θαλάσσι, θαλάσσια στα πλαίσια της Αταλάντα. Έχουμε καλό συντονισμό επιχειρησιακά, τοπικά και προσπαθούμε να βασιστούμε σε αυτήν τη συνεργασία και το συντονισμό ε, γιατί όπως ξέρετε η καταπολέμηση της πειρατείας δεν γίνεται μόνο στη θάλασσα αλλά γίνεται και στην ξηρά και έχουμε αυξήσει αυτή τη συνεργασία με την Κίνα. Με συνεργασία στην Ξηρά, ε, για, στη Σομαλία και στο κέρας Αφρικής εν γέννη. Μία άλλη περιοχή, ένα τομέα που πρέπει να συνεργαστούμε και το προσπαθούμε, είναι εκεί όπου έχουμε ειρηνευτικές αποστολές. Μαλή, προφανώς είναι υποψήφια χώρα, προφανώς. Προσπαθούμε πολύ έχουν γίνει συνεδριάσεις μεταξύ των διοικητών και των δύο πλευρών και καταρτίζουμε ένα κατάλογο δράσεων που θα μπορούσαμε να κάνουμε και προς, έκπληξή μου δεν δόθηκε συνέχεια από την Κίνα ε, μέχρι στιγμής ε, γιατί η συνάντηση αυτή έγινε πριν από ένα χρόνο και πλέον Επίσης γίνονται σεμινάρια υψηλού επίπεδου για την ασφάλεια και την άμυνα. Η κατάρτιση είναι καλή, ξεκινάμε από χαμηλό επίπεδο. Ε, η γνώση του ενός για τον άλλον είναι πολύ σημαντική. Προσκαλούμε ε, μεσαία στελέχη και ανώτατα στελέχη, αξιωματούχους, στρατιωτικούς να συμμετάσχουν σε αυτά τα σεμινάρια και συνήθως εκεί εξηγούμε την ΚΠΑ που συχνά εντυπωσιάζει τους συνομιλητές μας. πρέπει να πούμε πολλά για να εξηγήσουμε τις λειτουργίες, έστω και με σχηματικό τρόπο της ΚΠΑ. Αλλά το να βασιστούμε σε μια επιτυχημένη αποστολή όπως η Αταλάντα είναι σημαντικό ε, και βοηθάει. Υπάρχουν και άλλες ιδέες που δεν ήταν τόσο επιτυχής. Κάποια στιγμή ε, είχαμε μια κοινή άσκηση κατά πολέμης της πειρατείας Θέλουμε τέτοιες ασκήσεις να τις πολλαπλασιάσουμε, αλλά αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Έχουμε προσκαλέσει τον Κινέζο Υπουργό Άμυνας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε τις επαφές στρατιωτικών Κινέζων και Ευρωπαίων στις Βρυξέλλες, στο Πεκίνο, στους τομείς όπου υπάρχουν και επιχειρήσει επιχειρήσεις, μπορούν να υπάρξουν νέε επιχειρήσει π.χ. Μαλή. Ελπίζω επίσης να υπάρχει υψηλότερη δέσμευση από τους Κινέζους ε, σε ευθεία γραμμή με την αυξανόμενη οικονομική ισχύ της ε, Κίνας ε, που θα μπορούσαν να συνοδεύσουν νιοπομπές αποστολής τροφίμων αλλά τελευταία ήταν πριν από ένα-δύο χρόνια. Για το 16 1. Υπάρχει μια διμερής διάσταση ε, που είναι χρήσιμη για τους 11. Έρχονται, έχει έρθει ο Πρωθυπουργός της Κίνας. Επιτρέπεται να έχουμε διμερείς σχέση, έτσι. Ε, υπάρχει μια διάσταση ε, η οποία όμως είναι ανησυχητική εκεί το 16-1 στην αρχή ε, ήθελε να εφαρμόσει το BOR, το μία ζώνη, μία, ένας δρόμος. Αλλά αυτό ήταν διέξοδο, γιατί η κινέζικη προσφορά δεν είναι ανταγωνιστική. Εκτός κι αν είσαι από συγκεκριμένες χώρες, όπου ψάχνεις να βρεις οτιδήποτε για να πλήξεις τις Βρυξέλλες, ε, εάν δεν είσαι από τη συγκεκριμένη χώρα που είσαι εντελώ, που Αλλεργίε στι Βρυξέλλε, α πούμε. Αλλιώ, αν προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη χώρα από, από αυτέ, ε, δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Ε, υπάρχουν ε, πολλαπλέ, υπερβολικά πολλέ συνεδριάσει υπουργών κτλ. Ε, τώρα δεν θέλω να συζητάνε πια τι υποδομέ. Συζητούν ε, διάφορε δράσει σε τομεί όπου έχουμε ήδη συνεργασία με την Κίνα. Υπάρχει και η υποπεριφερειακή διάσταση που μας ανησυχεί. Παρακολουθούμε του συνεγγύς και αυτό το επίπεδο, αλλά συνεργαζόμαστε σε κάποια επίπεδα. Ε, δεν μας αρέσει το 16 αλλά δεν μας προσκαλούν οι Κινέζοι στο επίσημο κομμάτι της συνεργασίας. Για την Ταϊβάν Ε, να σας πω ότι ε, θέλω να διορθώσω κάτι που είπα ε, για τον ΠΟΗ, όχι τον Οργανισμό των Ομοίων. εδώ προσπαθούμε να βοηθήσουμε την Ταϊβάν. Ε, έρχομαι σε επαφή με κράτη-μέλη που έχουν ίδια νοοτροπία, ίδια άποψη. Δεν τα βλέπει ο κόσμος αυτά, δεν τα ξέρει ενδεχομένως. Ε, για την εικόνα 501, αυτό είναι ακόμα ένα παράδειγμα για να αυξήσει εκείνα την πίεση της στην Ταϊβάν. Η Ταϊβάν δεν ανήκει σε κανένα φορέα αεροπορίας, σε καμία οργάνωση αεροπορίας. Υπάρχουν μόνο διμερείς συμφωνίες μεταξύ των δύο και οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπαίνουν στον αεροχώρο που ελέγχει τα Ιβάν. Αναγνωρίζεται η διάσταση της ασφάλειας από εμά, Ε, γιατί μην ξεχνάτε ότι θα μπορούσαν πίσω από τα πολιτικά αεροσκάφη να κρύβονται στρατιωτικά αεροσκάφη. Πάντως ε, σημείωσα την άποψη της πλειοψηφία ότι θα έπρεπε εδώ να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προς το παρόν δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτά νομίζω ότι αρκούν τα όσα είπα. Η κυρία Πέισοβα, η επόμενη μιλητρία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Κρίστοφ Μανέ. Για το ζήτημα της Ταϊβάν είναι πράγματι πολύ δύσκολο το θέμα αυτό. Αλλά βεβαίως όπως και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς τα περιθώρια διεθνούς δράσης είναι πάρα πολύ περιορισμένα και αυτό αφορά βέβαια και την Ευρώπη. Όσον αφορά ε, την, την ασφάλεια, αυτό είναι προφανώς ένα από τα θέματα. Κατά τη γνώμη του Πεκίνου όμως πρόκειται για εσωτερική τους υπόθεση. Άρα επαναρχόμαστε στην, στο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε. Πάντοτε αυτή είναι η κατάσταση σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Ταϊβάν. Υποθέτω ότι με κάποιον τρόπο τελικά τα θέματα αυτά θα διευθετηθούν σε διμερές επίπεδο. Και κάτι που στο τέλος θα παρουσιαστεί στον υπόλοιπο κόσμο ως μεγαλοψυχία του Πεκίνου. Κάτι τέτοιο θα συμβεί και στην, κατά πάσα πιθανότητα στη θάλασσα ε, της Ανατολικής Κίνας που ήταν ξεκάθαρα μια μονομερής ενέργεια αυτό που συνέβη, το περιστατικό αυτό στην, της Κίνας. Ε, άρα πρόκειται στην ουσία για ένα σημάδι από, την, από το Πεκίνο ότι καθόλου δεν προτίθεται να χάσει τον έλεγχο επί της Ταϊπέη το αντίθετο. Γι' αυτό και υπάρχει μια συνεχής κινητικότητα. Κάποιοι μάλιστα, εκεί στην περιοχή, κάποιοι μάλιστα λένε ότι η Ταϊβάν θα ήταν το ιδανικότερο δώρο για τα 100 χρόνια του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κάτι που είναι βεβαίως πολύ ανησυχητικό. και εντείνει ακριβώς και τις, τις ανησυχίες μας όσον αφορά την ασφάλεια. Αλλά ξέρετε, οι, οι, οι νομικές ε, συμβάσεις με την Κίνα, αν δεν, αν περιλαμβάνουν και μηχανισμούς επιβολής, δεν έχουν ε, ποτέ και ιδιαίτερη χρησιμότητα ή αποτελεσματικότητα. Ο Jinping και η Κίνα γνωρίζουν πολύ καλά ότι η πρώτη τους προτεραιότητα είναι η εσωτερική ασφάλεια και γι' αυτό και επενδύουν τόσο πολλά χρήματα σε, στο περιβάλλον, στην υγεία, στην ασφάλεια των τροφίμων. Ο προφανής στόχος όλων αυτών των κινήσεων είναι να εξασφαλιστεί η επιβίωση του ίδιου κόμματο. Αυτός είναι ο απότερο στόχος. Ε, είναι και μια κίνηση και μια μέθοδος ε, προκειμένου να, μπορούν, να μπορεί ο κινέζικος λαός να καταπιεί ευκολότερα τον απολυταρχικό χαρακτήρα του, του καθεστώτος. Δεδομένα για την κινέζικη άμυνα. Δεν θυμάμαι ποιος έθεσε αυτό το ερώτημα, αλλά το Σύπρι WWS, μια σειρά από φορείς έχουν διάφορα στοιχεία που αφορούν και την έρευνα και την, και την άμυνα. Ε, σχετική ε, μελέτη εκπώνησε και δημοσίευσε και ε, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας πρόσφατα ε, εδώ στο Residence Palace στις Βρυξέλλες μας θα παρουσιαστεί και επίσημα την Παρασκευή η σχετική μελέτη. Και τέλος, για το ερώτημα που αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Βεβαίω, δεν έχουμε περιθώρια να παρέμβουμε στα ζητήματα που άπτονται τις, ε, τα, εσωτερικά ζητήματα της Κίνας, όμως μπορούμε να επηρεάσουμε την ε, στάση της χώρας αυτής στα διεθνή φόρα. Ε, είτε μέσω της UNCLOS, είτε της ICA, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε στο να υπάρχουν συστήματα και μηχανισμοί που βασίζονται σε συγκεκριμένους κανόνες, αλλά ενδεχομένως εδώ στην περίπτωση της Κίνας να χρειάζεται λίγη περισσότερη προσπάθεια. Επίσης χρειάζεται να ενισχυθούν οι σχέσεις μας με την Κίνα. Πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι περισσότερο τους προσκαλούμε εμείς παρά εμείς εκείνοι, ε, εκείνοι εμάς. Υπάρχει βεβαίω και το ζήτημα για τα λιμάνια. Ε, αναφέρθηκε το, το λιμάνι ε, ε, ε στη Χαμπαντότα, αλλά ο Πειραιάς είναι απολύτως ευρωπαϊκό λιμάνι, άρα έχουμε κάθε λόγο να προσπαθήσουμε να ε, προστατεύσουμε και να εξασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα μέσω των ευρωπαϊκών υποδομών. Και εδώ μιλούμε για μεταφορές, για επικοινωνίες, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Ε, είναι ένα ε, πανευρωπαϊκό μάλλον πρόβλημα. Όταν για παράδειγμα στη Γαλλία εθνικοποιήθηκαν τα ναυπηγεία του Σαναζέρ ήταν, προηγήθηκε μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα σε κάθε περίπτωση αξίζει να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το θέμα να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι στρατηγικές μας προτεραιότητες να τις εξασφαλίσουμε μετά ε, σε δεύτερο επίπεδο ε, στη Χαμπαντόρτα οι Κινέζοι είναι, σίγουρα, ε, είναι σίγουρο ότι είχαν κάνει επενδύσεις προτού η Κόσκο αγοράσει το συγκεκριμένο ε, λιμάνι. λιμάνι. 16-1. Υπάρχει και σε υποπεριφερειακό επίπεδο το πρόβλημα αυτό. η Κίνα έχει καταβάλει προσπάθεια προκειμένου να ε, ενισχύσει την ε, επιρροή της και στην Μεσόγειο και στη Σκανδιναβία. Δεν συζητιέται πολύ συχνά αυτό το θέμα, αλλά πολύ, πολύ συχνά ε, δεν ξέρουμε αν πρόκειται για υπονόμευση Τη πολιτική τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια Ευρώπη, μια ενιαία φωνή, αν είναι διέρη και βασίλευε, ε, αν πράγματι, ή αν από την άλλη μεριά αποτελεί απλά μια κίνηση εξασφάλιση προστασίας των οικονομικών του συμφερόντων, ε, αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε κυρία Πέσοβα. Λυπάμαι, αλλά έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο και ήθελα να δώσω και το λόγο και στο τελευταίο μέλος του πάνελ για να μας πει δύο λόγια, οπότε ζητώ πολύ συγγνώμη που σας διέκοψα. Κύριε Σκόμπελ, ευχαριστώ απλά θα απαντήσω σε μια ερώτηση και θα κάνω ένα σχόλιο. Η ερώτηση, αν την κατάλαβα καλά, ήταν αν έχει αμυντική στρατιωτική στρατηγική η Κίνα και η απάντηση είναι ναι, αλλά, αλλά επίσημα για να ξαναπάμε σε ένα από τα έγγραφα κλειδιά που είναι η Λευκή Βίβλος για την άμυνα της Κίνας και αφορά ε, στρατηγική στρατηγική και εστιάζεται συγκεκριμένα σε αυτό το θέμα. Εκεί λέει η Κίνα ότι έχει ως στρα... Ε, στρατηγική στρατιωτική την ενεργό άμυνα. Ουσιαστικά είναι μια βασική στρατηγική αρχή αυτή η ενεργός άμυνα. Ε, μας πάει χρόνια πίσω τι λέει επίσης η Κίνα στο έγγραφο αυτό ότι είναι στρατηγικά αμυντική αλλά έτοιμη επιχειρησιακά. Οπότε αυτό σίγουρα ε, αποτελεί μια βασική έννοια. Έχω κάνει πολλές έρευνες για αυτό το θέμα. Έχω ψάξει να βρω διάφορα έγγραφα, αναλύσεις, ερμηνείες και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι η έννοια αυτή φαίνεται να καθιστά ασαφή τη διάκριση μεταξύ επίθεσης και άμυνας. Κάθε χώρα θεωρεί ότι πολεμά για να αμυνθεί. Ας είμαστε ειλικρινείς. Αλλά έχω διαβάσει ένα ολόκληρο βιβλίο γι' αυτό και δεν σας κουράσω τώρα με τις λεπτομέρειες. Αυτό αποτελεί πρόβλημα στην περίπτωση της Κίνας. Η Κίνα έχει αυτό που ονομάζω εγώ την οτροπία του συνοικού τείχους. Δηλαδή πάντα θεωρεί ότι δρά αμυντικά, ωστόσο δρά επιθετικά κατά περίπτωση. Αν δείτε τις επίσημες περιγραφές ε, της χρήσης στρατικών δυνάμεων από το 1949 από την Κίνα, παντού αυτές ονομάζονται ε, αντιπιθέσεις αυτοάμυνας. οι εμπειρογνώμονε μπορεί να διαφωνούν και να συζητούν ε, επόριστον κατά πόσο αυτό έχει νόημα ή όχι. Και η, η εισβολή στο Βιετνάμ το 1979, το ανατολούμε αυτό, αντιπίθεση αυτοάμυνα, ε, είναι κατάχρηση τη ορολογία ουσιαστικά. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Οι Κινέζοι είναι πολύ ειλικρινεί. Θεωρούν ότι είναι αμυντική δύναμη θεωρούν ότι υπεραμείνονται των δικών του συμφερόντων. Το πρόβλημα είναι ότι τα συμφέροντά του είναι επεκτατικά σε ολόκληρο τον κόσμο και στην περιοχή ε, και αποκτούν όλο και μεγαλύτερη δύναμη. Οπότε ο τρόπο με τον οποίο αυτό ερμηνεύεται, ο τρόπο με τον οποίο εκείνα βλέπει τη δική τη στρατηγική μα δημιουργεί ανησυχία. Ένα σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι σχεδόν όλοι όσοι γνωρίζω που μελετούν το Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό έχουν εκπλαγεί από το πόσο είναι η ταχύτητα του εξυγχρονισμού του στρατού και το πόσο γρήγορα έχει αποκτήσει νέες δυνατότητες σε οπλικά συστήματα ο Κινέζικος στρατός. Κινούνται πολύ ταχύτερα από ό,τι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος και οι περισσότεροι αναλυτές, από ό,τι είχαν πιστέψει. Και αυτό είναι σημαντικό. Στις παρατηρήσεις μου δεν ήθελα να υποτιμήσω τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά λόγω του εξυγχρονισμού του στρατιωτικού από την Κίνα ε, δημιουργεί προβλήματα στους γείτονές τους και ουσιαστικά σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεδομένων αυτών όμως ε, όταν αναφέρθηκα στα μέσα ε, της δεκαετίας του 2020 Πιστεύω ότι είναι σημαντική χρονική στιγμή που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Όπως ανέφεραν οι συναδέλφοί μου εδώ στο πάνελ, ο στρατός της Κίνας ε, ε, υφίσταται αυτή τη στιγμή μια ριζική μεταρρύθμιση. Τεράστιες αλλαγές ε, που συγκρίνονται με αυτές τον είπα πριν μερικά χρόνια. Δεν θα γίνουν ε, μια ανοιχτή αυτές οι αλλαγέ, ε, θα πάρουν χρόνια. Αυτή τη στιγμή ε, γίνονται τεράστιες οργανωτικές αλλαγέ στον PLA, αλλά σε 6-7 χρόνια από τώρα μπορεί κανείς να φανταστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα έχουν υλοποιηθεί πλέον και ο κινέζικος στρατός, ε, οι κινέζικες ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να λειτουργήσουν πλέον σε αυτό το νέο σύστημα. Οπότε αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το χρονικό πλαίσιο. Ε, έτσι, ε, βάσει αυτού θα πρέπει να ασχοληθούμε για να δούμε πού θα βρίσκεται η Κίνα στρατιωτικά σε εκείνη την εποχή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σκόμπελ. Συνάδελφοι, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε τη συνεδρίαση γιατί ορισμένοι από εμάς πρέπει να πάμε να συζητήσουμε το Brexit ε, με την ε, ε, Επιτροπή για το Brexit. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα διακεκριμένα μέλη του πάνελ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να στους χειροκροτήσουμε. Thank you.